Um, Καλημέρα σας. Ως συνήθως θα ήθελα καταρχήν να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Εγκρίνεται λοιπόν. Τα πρακτικά της 4ης Φεβρουαρίου εγκρίνονται. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Άρα εγκρίνονται. Οι ανακοινώσει του Προεδρείου θα γίνουν αργότερα αφού τελειώσει η συζήτηση με τους υπουργούς και πριν τις ψηφοφορίες. Λοιπόν, τώρα περνάμε στην ανταλλαγή απόψεων για τις προοπτικές της ένταξη της Λετωνίας στο ευρώ, στην Ευρωζώνη. Έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Κεντρικής Τραπέζης της Λετωνίας. Δεν ξέρω αν τα ονόματά σας μπορώ να τα προφέρω σωστά, αλλά όπως είπατε θα μιλήσει ο καθένας κατά πέντε περίπου λεπτά και μετά θα υπάρξουν ερωταπαντήσεις. Ποιος θα μιλήσει πρώτος? Εγώ. Εντάξει. Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Είμαι ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Λετωνίας και είναι μεγάλη μου χαρά μπορώ σήμερα να σας μιλήσω στις Βρυξέλλες. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές ε, της συνάντησης αυτής και όσους μας κάλεσαν εδώ πέρα σήμερα να εκφράσουμε τις απόψεις μας για τη Λετωνία να σας πω λίγα λόγια για τα οικονομικά της Λετωνίας. Πριν από 10 χρόνια ακριβώς ήταν η πιο γρήγορα αντισώμενη οικονομία. Ε, μια οικονομία η οποία ετοιμαζόταν για την ένταξη. Και πολλοί Λετωνοί ονειρεύονταν επίσης ε, μεγαλύτερη ανάπτυξη, ψηλότερη ποιότητα ζωής ε, και το να καλύψουν το και ενώ Με το να μην ε, είμαστε εντός Ευρωζώνης και το να είμαστε εκτός το 2008, δυστυχώς ε, αναγκαστήκαμε να περάσουμε μια δύσκολη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Αλλά το σημαντικότερο είναι να δούμε το τι έκανε η Λετωνία για να ξεπεράσει αυτή την κρίση και το πώς τα κατάφερε. Αυτό νομίζω θα μελετηθεί από πολλούς ε, πανεπιστημιακούς από τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα οικονομικά. Θεωρώ πως πολλοί συνειδητοποίησαν πως τα πιο αποφασιστικά στοιχεία της ε, πολιτικής κυβέρνησης ήταν η ταχύτητα, η δέσμευση, η αλληλεγγύη και η συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Σήμερα η Λετωνία και πάλι είναι η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη οικονομία στην Ευρώπη για ε, δεύτερη συνεχή χρονιά και είναι ενδιαφέρον για μένα να σας αναφέρω πως σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνεται πως η Λετωνία θα συνεχίσει να είναι η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη οικονομία για πολλά χρόνια ακόμα. Αλλά αυτό που είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι πως ε, το νόμισμα της Λετωνίας έχει συνδεθεί ήδη από το 1993 με ένα ε, καλάθι ε, νομισμάτων από το 2005 έχει συνδεθεί με το ευρώ και υπήρχαν βέβαια διάφορες κρίσεις, διακυμάνσεις αλλά η Κεντρική Τράπεζα κατάφερε να κρατήσει τη σύνδεση αυτή της ισοτιμίας η οποία λειτουργήσε πάρα πολύ καλά για μια μικρή και ανοιχτή οικονομία που αποτέλεσε έναν πυλώνα σταθερότητας και αποτέλεσε ο κύριο νομισματικό μέσο με το οποίο υλοποιήσαμε την νομισματική μας πολιτική. Γι' αυτό σήμερα εδώ μιλώντας ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι λυπηρό για μένα το να σας μιλάω για τους ε, καιρούς που πέρασαν με αυτή την σύνδεση. Αλλά πιστεύουμε πως στο μέλλον με το να μην έχουμε εθνικό νόμισμα η Λετωνία θα μπορεί να έχει ακόμη πιο σταθερό νόμισμα και θα μπορεί να επιτύχει ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα και να αποφύγει την ε, κερδοσκοπία που αντιμετωπίζουν οι μικρές ανοιχτές οικονομίες σε καιρούς κρίσης. Η προσπάθειά μας για να γίνουμε μέλος της ΟΝΕ είναι μακροχρόνια, αλλά η κρίση αυτή μας βοήθησε να αντιληφθούμε την αξία και τα σημαντικότερα στοιχεία της οικονομικής και νομισματικής σταθερότητας. Γι' αυτό το ευρώ ήταν για μας ένας φάρος, ένα άστρο λαμπρό που μας οδηγούσε για να επιτύχουμε τα κριτήρια του Μάστριχτ για για να γίνει η προσαρμογή, για να είμαστε έτοιμοι για το 2014 και να ενταχθούμε στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Από τον Σεπτέμβριο του 2012 η Λετωνία εκπληρώνει όλα τα κριτήρια του Μάστριχτ. Οπότε ως ενδιαφέρες της Λετωνίας ε, και για την εκπλήρωση των κριτηρίων νομίζω πως μπορούμε να μιλήσουμε ε, για αυτά τα ζητήματα αν θέλετε επιμακρών. Το σημαντικότερο είναι πως ε, είναι βιώσιμη η εκπλήρωση των κριτηρίων αυτή τη στιγμή είναι σε ιστορικό χαμηλό πληθωρισμός και έτσι θα παραμείνει. Είναι σημαντικό νομίζω να αναφέρω πως δεν είναι τυχαία η εκπλήρωση των κριτηρίων ε, αυτών ούτε είναι μόνο κάτι το πρόθεσμο και θα δημιουργηθούν προβλήματα στο μέλλον. Νομίζω πως η τελευταία κρίση ήταν τόσο έντονη που θα χαραχθεί στο μυαλό των Λετωνών για γενιές. Γι' αυτό πάρα πολλοί συνειδητοποίησαν το τι σημαίνει να ζούμε με τις δυνάμεις μας, ε, τι σημαίνει να έχουμε χαμηλό πληθωρισμό, να έχουμε παραγωγικότητα ε, που είναι συνδεδεμένη με την αύξηση των μισθών. Και αντιστρόφως, η αύξηση των μισθών πρέπει να συνδέεται με την παραγωγικότητα. τι θα αποκομίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Οικονομική και Νομισματική Ένωση από την ένταξη της ε, Λετωνίας. Θα το έλεγα περισσότερη Ευρώπη με το να ενταχθεί στην ΩΝΕ η Λετωνία νομίζω πως ε, θα μπορέσουμε να μοιραστούμε και εμείς τις εμπειρίες μας ε, σε καιρούς κρίσης και θα μπορούμε να συζητήσουμε τις διακυμάνσεις και τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που είχαμε και το δεύτερο πολύ σημαντικό νομίζω είναι πως όλοι θα δουν πως ε, η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση είναι ένα μεγάλο και στιβαρό πλοίο ε, στο οποίο θέλει να ανέβει και η Λετωνία και νομίζω τα χειρότερα πέρασαν. Επίσης θεωρούμε πως το κλίμα είναι σωστό, υπάρχει στήριξη, υπάρχουν φίλοι που αναμένουν την ένταξη της Λετωνίας και άρα μια που είναι κατάλληλη στιγμή νομίζω πως η κυβέρνηση της Λετωνίας θα υποβάλει το αίτημα για την έκθεση σύγκλησης την επόμενη εβδομάδα και χαίρομαι για το ότι μπορώ να δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό για να εξηγήσει λίγο την ε, δημοσιονομική μας πολιτική. Καλημέρα σας κύριε και κύριοι. Η περίπτωση της Λετωνίας υπόσχεται πολλά, είναι πολλά υποσχόμενη. Πριν από μερικά χρόνια επλήγει από σοβαρή κρίση και έχασε σχεδόν 21% του ΑΕΠ της ξαφνικά. Μέσα σε 1,5 χρόνο έγινε αυτή η πτώση και αντιμετωπίσαμε πολλές προκλήσεις. Καταφέραμε όμως να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες και με τη βοήθεια και του Δουνουτού πετύχαμε αρκετά πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι expected είναι να αντιμετωπίσουμε τις δανειοληπτικές μας ανάγκες από τις αγορές. Ε, είμαστε, έχουμε εμπιστοσύνη ότι και στα επόμενα χρόνια η ανάπτυξή μας δεν θα είναι ασήμαντη. Εγκρίναμε το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας, το Fiscal Compact και προγραμματίσαμε για τα επόμενα χρόνια την ανάπτυξή μας, πράγμα το οποίο δεν θα μπορεί να γνωρίσει καμία επόμενη κυβέρνηση. Επίσης, καταφέραμε να συνδυάσουμε τα μέτρα λιτότητας με την αναδιάρθρωση της οικονομίας μας και τις μεταρρυθμίσεις που ήταν απαραίτητες. Πολύ καλός ο συνδυασμός γιατί η φρόνιμη δημοσιονομική πολιτική δεν απέκλεισε την ανάπτυξη. Γι' αυτό η Λετωνία μπορεί να προσβλέπει στο μέλλον με εμπιστοσύνη. Και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και οι επιχειρηματίες δείχνουν την ίδια εμπιστοσύνη. <clears throat> Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι πώς να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην παιδεία, στον υγειονομικό τομέα, στην εργασιακή πολιτική. όλο και πλησιάζουμε σε εξισορρόπηση του προϋπολογισμού μας και αναμένουμε πρωτογενή πλεονάσματα για να μπορέσουμε να διαθέσουμε περισσότερα χρήματα σε απαραίτητα προγράμματα που τα εγκρίνει και η Κομισιόν και το Δουνουτού. όπως τη μείωση των ανισοτήτων και της ανέχειας και αυτή τη στιγμή ήδη προγραμματίζουμε για του χρόνου αυξήσεις του κατώτατου μισθού και ορισμένων φόρων για πιο δίκαια φορολόγηση. Αυτό είναι κατανοητό γιατί υπήρξε η κρίση αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερα έσοδα και γι' αυτό μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά τα μέτρα. Πράγματι πιο πολύ σημαντικά είναι όλα αυτά και για άλλα έθνη να μπορέσουν δηλαδή να συνδυάσουν την δημοσιονομική φρόνηση με μεταρρυθμίσεις που να μην αποκλείουν την ανάπτυξη. Αυτό το έχει αποδείξει η Λετωνία. η Λετωνία νομίζω έχει λύσει πια το πρόβλημα. Αλλά ξέρουμε ότι η κρίση της Ευρωζώνης δεν έχει τελειώσει συνολικά. Και οι βαλτικές χώρες όμως πήραν μέτρα ανάλογα, οι υπόλοιπε βαλτικές χώρες ανάλογα με τις Λετωνίας και μπορεί να αποτελέσουν όλα αυτά παράδειγμα για την λήψη των αποτελεσματικότερων μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης. Επίσης πολύ σημαντικό είναι νομίζω ότι η χώρα μπαίνοντας στην Ευρωζώνη θα φέρει σε αυτήν μία νέα προοπτική. Πράγμα το οποίο είναι σημαντικό για όλη την Ευρώπη. Εμείς είμαστε πάντως αποφασισμένοι να ενταχθούμε στο ευρώ, πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν μπόρεσε να γίνει μέχρι τώρα. Τώρα όμως με τα στοιχεία αυτά που σας ανέφερα δημοσιονομικής φρονήσεως και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία μας, η χώρα είναι έτοιμη να ενταχθεί στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως τα γνωρίζετε όλοι, η κυβέρνηση της Λετωνίας μας είπε ότι πρέπει, ε, μάλλον πρέπει να αναφέρεται σε εμά ε, και στο, Συμβούλιο και στην Κομισιόν σε σχέση με τον προ, την πρόοδο της χώρας ως προς την επιτυχή υιοθέτηση του ευρώ. Και έπειτα η Κομισιόν θα φτιάξει μια ανέκθεση ε, την την Άνοιξη. Εμείς έχουμε ήδη ορίσει εισηγητή για την έκθεση αυτή και είναι ο κύριος Μπόλτς, Μπέρκαρτ Μπόλτς. Και μπορείς να πάρεις το λόγο για την πρώτη ερώτηση, Μπέρκχαρτ. Το φόρματ που χρησιμοποιούμε είναι ότι έχουμε χρονοθυρίδα 5 λεπτών για ερωταπαντήσεις και θα αφήσω στους προσκεκλισμένους μας να επιλέξουν ποιες ερωτήσεις θα απαντήσουν για να μην μπορεί να υπάρξουν δύο απαντήσεις ας πούμε σε κάθε περίοδο. Ναι, ευχαριστώ κυρία Υπουργέ κύριε Υπουργέ, κύριε Διοικητά. Χαίρομαι για το ότι ήρθατε εδώ πέρα για να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση για τα ουσιαστικά ζητήματα, για την ε, προσχώρηση της Λετωνίας στην Ευρωζώνη. Εγώ χαιρετίζω τη φιλοδοξία της Λετωνίας να ενταχθεί στο ευρώ τον Ιανουάριο του 2014. Νομίζω πως είναι ένα εξαιρετικά καλό παράδειγμα για την εξυγίανση του προπολογισμού και την επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης χρέους. Και ακριβώς ε, σε αυτή τη στιγμή η θέληση της Λετωνίας να ενταχθεί στο ευρώ νομίζω πως είναι ένα πάρα πολύ καλό μήνυμα εμπιστοσύνης ε, στο νόμισμά μας και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα εστιαστώ σε λίγα πράγματα. Για μένα το πρώτο σημαντικό ερώτημα είναι πώς ε, βγήκε από την κρίση η Λετωνία, πώς ε, αντιμετώπισε την κρίση χρέους, τι μπορούν πιθανώς να μάθουν ε, άλλα κράτη-μέλη που είναι ήδη στην Ευρωζώνη από την Λετωνία. Μετά. Με ενδιαφέρει να μάθω ποια συγκεκριμένα μέτρα ελήφθησαν για να διασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών Κατόπιν ένα ερώτημα για τον πληθωρισμό. Πόσο σίγουροι είστε πως ε, ο πληθωρισμός ε, είναι υπό ε, υποέλεγχο. Τελευταίο που με ενδιαφέρει υπάρχουν βεβαίως διαφορές εκθέσεις, αλλά αποφασιστικό είναι ε, να θέλει και ο λαός αυτή, αυτό το βήμα προς την Ευρωζώνη και σε σας ε, ε, νομίζω υπάρχει αίσθηση πως η χώρα είναι ακόμα αναποφάσιστη. Υπάρχει κάποια θετική τάση αποδίδουν οι καμπάνιες οι οποίες γίνονται για το ευρώ. Αυτά θα ήθελα να σα ρωτήσω. Ευχαριστώ. Πολλέ ερωτήσεις για να απαντηθούν σε δυόμιση λεπτά. Οπωσδήποτε θα ακουστούν ε, και θα απαντηθούν και μετά. Θα ξεκινήσω με το πώς αντιδράσαμε στην κρίση. Καταρχήν, διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να ενεργήσουμε γρήγορα και σωστά. Πολύ σημαντικό ήταν το ότι δημιουργήσαμε ε, εξ αρχής ε, κοινωνικό διάλογο από την αρχή της κρίσης. Και επίσης ε, φτιάξαμε μια ομάδα διαχείρισης των μεταρρυθμίσεων που εξακολουθεί να υπάρχει. Κυβέρνηση, συνδικάτα και επιχειρηματίες ανταποκρίθηκαν και ε, εξετάσαμε όλα τα μέτρα λιτότητας, οποιαδήποτε πρόταση, πρόταση μεταρρύθμισης. Αυτή τη στιγμή ε, εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με, με όλα αυτά τα θέματα. Διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να γίνουν περισσότερα και γρηγορότερα. Ε, πρώιμη εφαρμογή είναι πάρα πολύ σημαντική, το front loading, ιδιαίτερα για τις μικρές χώρες. Εάν θέλεις να έχεις ε, και πάλι την εμπιστοσύνη της αγοράς, θα πρέπει να αντιδράσεις σωστά. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, η γρήγορη αυτή αντίδραση. Ταυτόχρονα καταφέραμε ε, και επιβιώσαμε δύο εκλογικές διαδικασίες και οι ψηφοφόροι στήριξαν την πολιτική λιτότητα γιατί Πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι και αλλά όχι αγνοώντας αυτές τις αλλαγές και την εξυγίανση. Τα μέτρα αντιστοιχούν στο 17% του ΑΕΠ, 17% του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια των 2-3 ετών. Τα 2 τρίτα από την πλευρά των δαπανών και το 1 τρίτο μόνο από την πλευρά των εσόδων. πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινάμε από την πρώτη-δεύτερη χρονιά για να κάνουμε ό,τι ε, μπορούμε καλύτερο. Ευχαριστώ. Τελείωσε ο χρόνος για τις συγκεκριμένες απαντήσεις. Εγώ θέλω να πω δύο λόγια παραπάνω ε, για την ερώτηση που αφορούσε την επιστροφή του πληθωρισμού. Πρέπει να αναφέρω νομίζω τρία στοιχεία. Όλοι σαφώς αναγνωρίζουν ότι οι μισθοί θα μπορούσαν να αυξηθούν μόνο όταν υπάρξει παραγωγικότητα. Και υπάρχει παραγωγικότητα. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό Τώρα, ο προϋπολογισμός. Οι Ευρωπαίοι και οι ε, Λετωνοί νομοθέτες έχουν ε, ε, εκπονήσει και ακόμα σκληρότερους προϋπολογισμούς από ότι πριν μάλλον να κάνει το Κοινοβούλιο προτείνει το εξαπλό πακέτο δεν, εφόσον υπάρχει ακόμα έλλειμμα στον προπολογισμό, δεν υπάρχει χώρος για επιπλέον συμπίεση των τιμών, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε ότι υπάρχει μόχλευση στον τομέα του τραπεζικό, που σημαίνει ότι ο δανεισμός δεν θα επανέλθει στο εγγύς μέλλον. Πράγμα το οποίο τελικά θα συμβαδίσει με την οικονομική ανάπτυξη. Όσον αφορά τη στήριξη του ευρώ, κάποιοι συνάδελφοι έχουν θεωρήσει πως είναι πολύ ψηλή η στήριξη δεδομένου το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο και σε κάποιες από τις χώρες. Νομίζω πως έχουμε μια πολύ άνετη κατάσταση όπου έχουμε το 30% υπέρ της Ευρώπης 30 περίπου κατά και, 30, και ακόμα 30 ή 35 που είναι αναποφάσιστοι. Είναι ο κατάλληλος χρόνος λοιπόν για να εξηγήσουμε περισσότερο, να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και έτσι να είμαστε πολύ ξεκάθαρα αποφασισμένοι ώστε να αυξήσουμε τη στήριξη για το ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ερώτηση από την Ελίζα Φερέιρα από την ομάδα των Σοσιαλιστών. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση, οι ερωτήσεις μου αφορούν την βιωσιμότητα της απόδοσης που φτάσατε. Διότι πιστεύω ότι αν τώρα δει κανεί την Ευρωζώνη και πώς λειτουργεί, το πρόβλημα είναι ε, η πραγματική οικονομία των κρατών μελών, πώς θα μπορέσει να ακολουθήσει τον δρόμο της ε, βιωσιμότητας. Εγώ ανησυχώ όχι μόνο για την ονομαστική σύγκληση, αλλά και για την βιωσιμότητα της πραγματικής σύγκλησης της οικονομίας. Όλος ιδιαίτερος θα ήθελα να δούμε τους λόγους για τους οποίους υπάρχει η μακροοικονομική ανισορροπία σε σχέση με το εξαπλό πακέτο. Σε σχέση με τη Λετωνία, εδώ βλέπουμε την ανεργία Ξέρω πως έχετε κάνει μεγάλες προσπάθειες, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω ποιες είναι οι προπτικές για την απασχόληση και την μετανάστευση. Και δεύτερον, ο ρόλος των, ε, της φορολόγησης και των, ε, των ξένων ε, άμεσων επενδύσεων. Πόσο εξαρτάται η χώρα από αυτό. Τώρα, ενιαίο αποπτικό σύστημα που δημιουργούμε για τις τράπεζες. Σε ποιο βαθμό η δομή του τραπεζικού συστήματος ιδιαίτερα σε σχέση με χώρες εκτός Ευρωζώνης ή που δεν θα μπουν στην Ευρωζώνη, πώς αυτό επηρεάζει τη θέση σας σε σχέση με τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Είναι πολύ σημαντικό για όλους να δείχνουν τη βιωσιμότητά τους για την ανάπτυξη. Αλλά δείτε τα στοιχεία ε, τα οποία ε, παρουσίασε η Λετωνία για το 2012-2013 μπορείτε να δείτε πως υπάρχει βιωσιμότητα και σταθερότητα των στοιχείων. Μπορούμε να δούμε ότι από το Σεπτέμβριο και έκτοτε πληρούμε όλα τα κριτήρια του Μάστρεχτ. Είναι ενδιαφέρουσα η κατάσταση γιατί διατηρείται η ταχύτερη ανάπτυξη και χαμηλότερος πληθωρισμός και στις προβλέψεις της Κομισιόν τα επόμενα 2-3 χρόνια σχεδόν τα ίδια παραμένουν τα στοιχεία, δηλαδή χαμηλός πληθωρισμός και σταθερή ανάπτυξη και γρηγορότερη. Όπως είπα αυτή τη στιγμή, είμαστε σε θέση να εστιάσουμε περισσότερο στις διαφορετικές ε, μορφές. Εμείς αλλάζουμε τη δομή της οικονομίας μας και έχουμε, πιστεύω, ένα πολύ καλό δυναμικό για τη βιομηχανία παραγωγική και εξαγωγική και έχουμε και την κατάλληλη υποδομή, γιατί ακόμα και τώρα έχουμε διψήφιο ποσοστό εξαγωγών. Οι επιχειρήσεις μας είναι πιο αποτελεσματικές, ο δημόσιος τομέας μας είναι πιο αποτελεσματικός και η εισαγωγή των μέσων που εμποδίζουν τις περιττές δαπάνες ε, είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Όπως σας είπα, η, η ανεργία μας συρρυκνώνεται στην ε, Λετωνία και σε ολόκληρη τη Βαλτική γρηγορότερα από ό,τι σε άλλες περιοχές και έχουμε, ε, έρθει, έχουμε κατέβει από το 17,3% της ανεργίας που ήταν στη, το, το ανώτερο μας ποσοστό στη χειρότερη περίοδο της κρίσης ε, έχουμε κατέβει λοιπόν στο 10% και στοχεύουμε να κατεβούμε σε μονοψήφιο νούμερο πριν το καλοκαίρι. Όπως σας είπα, στόχος είναι δύο πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Παιδεία, εκπαίδευση δηλαδή του εργατικού δυναμικού και ο άλλος δεύτερος στόχος αφορά την εργατική πολιτική, την πολιτική μάλλον απασχόλησης. Ε, έχουμε ε, χρόνο, όπως σας είπα, τα νούμερα για την ανεργία προχωρούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι. Anything to add or... I think there was a question about SSM. Έχετε κάτι να συμπληρώσετε, ναι, για τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας. Όπως θα ξέρετε, η Λετωνία αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχει σε αυτές τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Έχουμε, περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τη θέση μας Ωστόσο, η Λετωνία είναι έτοιμη να συνεργαστεί σε όλα τα μέτωπα και να προσχωρήσει στον μηχανισμό εποπτείας όσο γίνεται πιο σύντομα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Εξ της Άλτε, η Σιλβί Γκουλάρ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Διοικητά. Νομίζω ότι αν πληρείτε τα κριτήρια για την ένταξη στην Ευρωζώνη είναι πολύ καλό νέο για το μέλλον και το δικό σας και της Ένωσης ολόκληρης. Ευχαριστώ λοιπόν για όσα κάνατε, αλλά θα ήθελα επίσης να πω ότι <clears throat> βρισκόμαστε σε μεταβατική περίοδο. Πώς βλέπετε εσείς το ρόλο σας στο μέλλον. Υπάρχει τάση σήμερα να θεωρούμε ότι τα 17 μέλη της Ευρωζώνης είναι λίγα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης, αλλά ο μηχανισμός αυτός εποπτείας δεν θα λειτουργήσει παρά μόνο αν λάβουμε υπόψη και το ρόλο που θα παίξουν οι υποψήφιες χώρες για την Ευρωζώνη. Πρέπει δηλαδή μήπως να παραμείνει η διαίρεση αυτή μεταξύ των 10 και των 17 είναι σίγουρο ότι δεν θα παραμείνει. Εσείς πώς το βλέπετε λοιπόν στις διαπραγματεύσεις και πώς θα μπορούσατε να πείσετε ορισμένες χώρες ότι και όσες θα ενταχθούν, ε, ότι καμία δεν αποκλείεται, ότι και εκείνες μπορούν να ενταχθούν δηλαδή. Um, uh, Κοιτάξτε, με βάση την πρόσφατη εμπειρία της Λετωνίας βλέπουμε πολύ καλά, καταλαβαίνουμε σε ποια κατεύθυνση, προς πού πρέπει να κινηθεί η Ευρωζώνη και πώς να αλλάξει. Εμείς είμαστε υπέρ προτάσεων που θα φέρουν την Ευρώπη και την Ευρωζώνη σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Για μας είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα ως προς την εποπτεία των τραπεζών και τους υπόλοιπους μηχανισμούς. Τέτοιες προτάσεις τις υποστηρίζουμε. Γιατί έχουμε την πρόσφατη εμπειρία μας η οποία λειτουργήσε πολύ καλά και αποτελεσματικά και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από άλλες χώρες. Δεχόμαστε όλες τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν, όλες. Είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίζουμε πάντοτε δύο πράγματα. την τωρινή κατάσταση με τη μελλοντική. Σε αυτή την περίοδο τα τελευταία 5-6 χρόνια η Λετωνία έμαθε πολλά. Θα υπάρξουν πάρα πολλές συζητήσεις και μελέτες μεταξύ ακαδημαϊκών για την αξιολόγηση των μέτρων και για την αντιμετώπιση της κρίσης αλλά πιστέψτε μας έχουμε και εμείς μια πολύτιμη εμπειρία ρωτήστε μας και θα σας πούμε ναι μόλις σας ρώτησα αλλά δεν μου απαντήσατε λοιπόν το ερώτημά μου ήταν τι θα κάνετε τους επόμενους μήνες για το SSM τι θα κάνετε δεν γνώριζα καν ότι θα χρειαζόταν να πω κάτι για το SSM. Όταν θα έχουμε επιλογή μεταξύ α, β, γ θα σας απαντήσουμε, αλλά δεν θέλω να σας πω κάτι υπερβολικά γενικό το οποίο δεν θα έχει καμία επίπτωση. Ναι, δεν έχει τελειώσει ακόμα η ένταξή τους και στο SSM, δεν ξέρουν ακόμα τι θα κάνουν, γι' αυτό δεν απαντάει θα μπούμε, θα μπούμε. Αυτό δεν είναι αμφίβολο. Το θέμα είναι απλώς μετά τι θα γίνει. Προς τα πού θα κινηθούμε μετά. Τι πρόσθετα προβλήματα θα μας τεθούν από το SSM. Έχετε λοιπόν μια απάντηση. Θα μπουν στο SSM. I'm sorry, Sharon, but my question was ναι, αλλά για τον διαχωρισμό σε δύο τμήματα μεταξύ χωρών της Ευρωζώνης και μη χωρών της Ευρωζώνης ή χωρών της μη Ευρωζώνης, τι φρονείτε, οι υπόλοιπες χώρες θα θελήσουν να μπουν. Ναι, εμείς θα αποτελέσουμε γέφυρα. γιατί αντιμετωπίσαμε προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν ή αντιμετωπίζουν και οι άλλες φορές που δεν είναι στην Ευρωζώνη και οι οποίες μελετάνε πολύ προσεκτικά την εμπειρία μας. Η αποδοχή ενός τέτοιου μηχανισμού και από αυτές θα ήταν πολύ σημαντική και εμείς μπορούμε να αποτελέσουμε γέφυρα. έχουμε την εμπειρία μας και μπορεί να αποτελέσει για αυτές μάθημα. Για όσες δεν έχουν τουλάχιστον αποφασίσει να ενταχθούν στην Ευρωζώνη. Συνεννοούμαστε και μας ζητάνε και αυτές τις πληροφορίες. Και αυτό θα επηρεάσει, θα έχει επίπτωση σε όλες τις χώρες μέλη. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν το θέμα του χρόνου επόμενο ερώτημα των συντηρητικών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω κάτι. Ε, στο κόμμα μας δεν υπάρχουν πολλοί ευρωβουλευτές από τις χώρες της Ευρωζώνης και οι θέσεις μας γενικά ε, είναι πως δεν πιστεύουμε στο λαμπρό μέλλον της ε, Ευρωζώνης. Σεβόμαστε βεβαίως την πολιτική απόφαση να ενταχθούμε στην Ευρωζώνη και θα την στηρίξουμε. Τώρα, το να είναι κανείς πάνω στη γέφυρα δεν είναι και πολύ καλή θέση γιατί ή ανάμεσα σε δύο βάρκες θα έλεγα καλύτερα γιατί μπορεί να βρεθεί κανείς στο νερό. Γνωρίζουμε την ε, η ιστορία μας πως εδώ και 20 χρόνια ήμασταν ε, μια γέφυρα μεταξύ ισχυρών χωρών και η προσπάθειά μας να ενταχθούμε στη Δυτική Ευρώπη ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε, όπως είπα, η θέση αυτή είναι δύσκολη, αλλά για να έχουμε κάποιο όφελος για τους μελλοντικού μας εταίρους στην Ευρωζώνη, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφιβολία για την βιωσιμότητα των οικονομικών μεγεθών. Και γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε για κάποια ζητήματα τα οποία δεν είναι τελείως θετικά. Το ένα είναι η κοινωνική ανισότητα και θα ήθελα ο Υπουργός Οικονομικών να μας πει τι ε, μέτρα θα ληφθούν σε αυτό το μέτωπο γιατί πρέπει να υπάρχει βεβαίως και μια πολιτική βιωσιμότητα της πολιτικής μας. Έχουμε εκλογές ε, και θα... Ε, βεβαίως δεν εκλέγεται ο διοικητής κεντρικής τράπεζας, αλλά Έχουμε εκλογές. Πρέπει να δούμε το τι θα γίνει, γιατί είδατε και τι έγινε με τις πρόσφατες εκλογές στην Ιταλία. Το δεύτερο ερώτημα αφορά τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Όλοι αναμένουν μια, τη λύση στην Κύπρο, το τι θα γίνει θα μπορούσε να υπάρξει ένα κούρεμα των μεγάλων καταθέσεων από τρίτες χώρες ή χωρίς αυτό. Τι θα προτιμούσατε εσείς λαμβάνοντα υπόψη του τι θα είναι καλύτερο για το τραπεζικό τομέα της Λετωνίας ε, ε, αναλόγως και με το πώς θα εξελιχθεί η κρίση στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Όπως είπα, υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Είναι κορυφαία προτεραιότητα για τον προπολογισμό του επομένου έτους και ο Υπουργό Οικονομικών, εγώ δηλαδή και ο Υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας παρουσιάσαμε ένα σχέδιο και οι προτάσεις της ε, Κομισιόν και της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Δόνου του εξετάστηκαν και πρέπει βεβαίως να δούμε την ανισότητα. Τι θα κάνουμε λοιπόν του χρόνου. Θα αυξήσουμε τον ε, κατώτατο μισθό θα διπλασιάσουμε το ποσοστό, ποσό του ελάχιστου το ποσό στο οποίο επιβάλλεται η ελάχιστη φορολογία και βεβαίως ε, θα υπάρξει και ένα επίδομα για τα εξαρτώμενα άτομα γιατί βεβαίως ε, και στο δημογραφικό μέτωπο έχουμε αύξηση των ε, γεννήσεων και αυτό είναι σημαντικό γιατί είμαστε μια μικρή χώρα. Δηλαδή πώς θα μειώσουμε τη φτώχεια και πώς θα βοηθήσουμε τις οικογένειες. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Έχουμε περισσότερα φορολογικό έσοδα. Μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό και να απαντήσουμε με τις, με τις ε, πολύ σημαντικές αυτές ε, πολιτικές που ούτως ή άλλως αναμένει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Δούνου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό κάνουμε λοιπόν, αναψώμεθα και μειώνουμε την φτώχεια. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι δεσμεύσεις μας και έχει δεσμευτεί σε αυτό η κυβέρνηση. Ε, εγώ απόρρισα λίγο για το ερώτημά σας. Γνωρίζετε πως ε, η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο 31 Ιανουαρίου ενέκριναν ε, έναν νόμο ο οποίος ξεκάθαρα ορίζει πώς θα αλλάξουν ε, πώς θα αλλάξει το, το νόμισμα ότι δηλαδή θα είναι απεριόριστα τα ποσά για, για δύο μήνες και μετά για τρεις μήνες πρέπει να πάει κανείς σε τράπεζα και ταχυδρομείο όχι όχι μάλλον παρεξηγήσετε την ερώτησή μου ρώτησα το διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, γνωρίζουμε όλοι εδώ μέσα πως ε, κάπως θα βοηθηθεί η Κύπρος από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, από την Ευρωζώνη, από το δόνο για να λυθεί το, το πρόβλημα. Και από μεθοδολογική σκοπιά είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα λυθεί αυτό το ζήτημα. Με κούρεμα των μεγάλων καταθέσεων από τρίτες χώρες ή χωρίς. Και το ερώτημά μου, επειδή η Λετωνία θα ενταχθεί στην Ευρωζώνη, ελπίζουμε σε ένα χρόνο, όλοι ελπίζουν σε αυτήν την αίθουσα, ε, το ερώτημά μου είναι ποια είναι η προτίμησή σας για την, προτίμηση, για την ε, λύση που θα δοθεί στην Κύπρο. Να Λαμβάνοντας υπόψη και το τι συμφέρει την Λετωνία. Ε, υπενήσεστε πω όλοι εντός τη αίθουσα γνωρίζουν τα πάντα. Όχι, δεν γνωρίζουν όλα τα πάντα. Η κατάσταση είναι περίπλοκη και οπωσδήποτε δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα πει αν θα πρέπει να ακολουθηθεί μία κατεύθυνση ή η άλλη, ειδικά χωρίς να ξέρω όλες τις ε, επιπτώσεις ε, και τις δυσκολίες ε, που αντιμετωπίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου. Θα ήθελα να σχολιάσω πως οι διαδικασίες αυτές δεν είναι οπωσδήποτε διαφανείς για, για προφανείς λόγους. Και μια επιτυχία του Κοινοβουλίου ήταν πως τουλάχιστον το, τουλάχιστον το Προεδρείο θα έχει κάποιες εμπιστευτικές ενημερώσεις για το τι γίνεται στις χώρες του προγράμματος, χωρίς να μπορούμε βεβαίως πάλι να σας πούμε μετά. Λοιπόν, περνάμε στους πράσινους τώρα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε. Η Λετωνία φαίνεται να τηρεί τα νομικά και οικονομικά κριτήρια αυτή τη στιγμή για να προσχωρήσει στην ζώνη του ευρώ και χαιρόμαστε πραγματικά. Ωστόσο, ωστόσο το γενικότερο πλαίσιο ε, μας ανησυχεί κάπως και θα ήθελα να σας ε, θέσω τρεις ερωτήσεις. Η μία ήδη αναφέρθηκε είναι το πλαίσιο του γενικότερου σκεπτικισμού που φαίνεται να βασιλεύει στη χώρα σας, στον πληθυσμό της χώρας σας όσον αφορά την προσχώρηση στην Ευρωζώνη. Γνωρίζουμε πως δεν είστε η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει το σκεπτικισμό του πληθυσμού, τι σκοπεύετε να κάνετε συγκεκριμένα για να κινητοποιήσετε και να εμπλέξετε την, ε, τον πληθυσμό της Λετωνίας σε αυτή τη δικασία προσχώρησης, γιατί εάν δεν μπλακεί ο πληθυσμός, τα πράγματα δεν λειτουργούν μόνο με τεχνικά μέσα. Δεύτερη επιτυχή που μας ανησυχεί ακόμη περισσότερο είναι οι πληροφορίες που έχουμε για ένα κάποιο επίπεδο αδιαφάνειας τραπεζικής στη χώρα σας που η κυβέρνηση δηλαδή έχει φτιάξει μια στρατηγική μείωση των ποσοστών φορολόγησης για να ευνοήσει την προσέλκυση κεφαλαίων. Αυτή η πολιτική που φαίνεται να έχετε υιοθετήσει δεν θα ευνοήσει το φαινόμενο της φορολογικής διαφυγής και του ξεπλήματος χρήματος, ιδιαίτερα από προέλευσης του μεγάλου γείτονά σας. Και έπειτα τι γίνεται με τη φορολογική σας πολιτική. Τρίτο στοιχείο, δικαίως αναφέρεστε σε μια σημαντική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Όμως αυτή η οικονομική ανάπτυξη εν μέρη δεν ξεπερνά το φυσικό σας κεφάλαιο. Θέλω να μιλήσω για την πολιτική μαζικής ε, αποψήλωσης των δασών, της, βασικής, της, ε, της μαζικής υλοτόμησης που αν δεν σταματήσει θα έχει αρνητικέ συνέπειες στο ποσοστά ανάπτυξή σας. Αυτά ήθελα να μου πείτε λοιπόν ε, κύριοι και ελπίζω να με καθησυχάσετε. Uh, uh, uh. Κοιτάξτε, το θέμα της κοινή γνώμης. Δεν είναι μυστικό πως η Λετωνία είναι ανάμεσα στις πιο σκεπτικιστικές φόρες για όλα τα θέματα αυτά και όχι μόνο για το ευρώ. Αυτή τη στιγμή γίνεται επικοινωνία για την εισαγωγή του ευρώ ε, και υπάρχει αυξανόμενη στήριξη ε, πιθανότατα σε δύο μήνες θα είμαστε στο 50-50. Ε, η πρώτη, το πρώτο θέμα που ανησυχεί είναι η κατάσταση της Ευρωζώνης. Ε, τώρα έρχονται όλο ένα και πιο θετικά νέα από πολλές από τις χώρες της Ευρωζώνης και ο κόσμος κατά κάποιο τρόπο συνειδητοποιεί πως όλες αυτές οι χώρες κάνει τα ίδια που έκαναν οι Λετονοί και οι χώρες της Βαλτικής, διαρροτικές μεταρρυθμίσεις, ε, αλητότητα, εξυγένση κτλ. Περιμένουν λοιπόν τα αποτέλεσματα, βελτιώνεται η κατάσταση στις περισσότερες χώρες. Ένα άλλο θέμα που αφορά την ε, επιφυλακτικότητα είναι ε, ο πιθανός πληθωρισμός, αλλά και πάλι έχουμε περάσει πολύ καιρό και έχουμε δώσει επιχειρήματα στις γειτονικές μας χώρες που πρόσφατα έγιναν μέλη της Ένωσης. Ε, ο πληθωρισμός αυξήθηκε, αλλά αυτό μας ωφελεί εμάς γιατί Εμπιστευόμαστε πολύ την Εστονία ως χώρα. Το παράδειγμα είναι δίπλα μας και εμείς θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Το, το έκαναν και οι Φιλανδοί πριν από λίγα χρόνια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος τελικά είναι πραγματιστής περάσαμε δύο εκλογικές διαδικασίες. Ήταν πολύ δύσκολο να δούμε αν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, αλλά τελικά ο κόσμος συνειδητοποίησε πως είναι ένας πολύ σημαντικός στρατηγικός στόχος και κατάλαβαν γιατί τον επιδιώκουμε. Πιστεύω πως η υποστήριξη λοιπόν θα αυξάνεται και χάρη στα καλά νέα που έρχονται από την Ευρωζώνη. Υπάρχουν πολύ καλές προθέσεις, πολύ καλές πολιτικές που ακολουθούνται στις διάφορες χώρες της Ευρωζώνης εν γέννη πρέπει να συνεχίσουμε. Μπορώ να σας ρωτήσω ότι αν καταναλώνετε μεγάλο τμήμα των πενταλέπτου με τις ερωτήσεις, δεν μπορώ να δώσω περισσότερο χρόνο για τις απαντήσεις. Πέντε λεπτά. Ο Νικόλας Χοντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Δικητά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Επαναλαμβάνω ότι είμαι από την ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για να σας θυμίσω ότι στην ομάδα μας υπάρχει λετονός ευρωβουλευτής, ο κύριος Ρούμπιξ. Δεν μας λείπει κατά μία έννοια ενημέρωση. Επομένως αυτά που θα σας ρωτήσω είναι θέμα αξιολόγησης. Πώς θα αξιολογείτε εσείς. Και δεύτερο, σας προσθέτω τίμα από την Ελλάδα για να αντιληφθείτε το πνεύμα της άλλης πτυχής των ερωτήσεων. Το πρώτο ε, είναι επιλογή σας αν θα μπείτε στο ευρώ. Είναι δικό σας θέμα. Το ερώτημα τίθεται σχετικά με την κοινή γνώμη και με τον κόσμο. Πώς θα το λύσετε αυτό το πρόβλημα. Ή θα ακολουθηθεί αυτό που λέει ο κύριος Όλι Ρεν, ότι για την περίπτωση της εισόδου στην Ευρωζώνη δεν λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο τι λένε οι πολίτες. Δώστε μου πιο σαφή απάντηση, δηλαδή πώς θα το λύσετε αυτό το θέμα. Δεύτερο, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, σας είπα για ποιο λόγο. Μου φαίνεται παράδοξο, οικονομικά και κοινωνικά παράδοξο, σε αυτή την περίοδο που η Ευρωζώνη έχει κρίση. Δεν ξέρω τι θετικά μηνύματα έχετε. Δεν ξέρω τι θετικά μηνύματα έχετε. Σας συνιστώ να μελετήσετε την εμπειρία και της δικής μου της χώρας και να μου δώσετε μια απάντηση τι προσδοκάτε σε σχέση με τα, τα στοιχεία της πραγματικής οικονομίας τα οποία αποφύγατε να αναφέρετε. Ανεργία, ανεργία των νέων, ε, κάτω από το όριο της φτώχειας ένα ποσοστό πληθυσμού. Άκουσα προθέσεις ότι θέλετε να τα αντιμετωπίσετε, σας το εύχομαι, αλλά η εμπειρία δείχνει ότι η Ευρωζώνη σήμερα δεν είναι τέτοια που να μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα. Και η τελευταία ερώτηση, επειδή άπτεται αυτού του ζητήματος, είπε ο κύριος ε, διοικητής της τράπεζας ότι το 2008 περάσαμε μια κρίση γιατί δεν είμαστε στην Ευρωζώνη. Διευκρινίστε μου σας παρακαλώ τι εννοείτε αν είσαστε στην Ευρωζώνη ήσασταν, θα είχατε τις δυσκολίες δανεισμού που είχε και η δική μου χώρα και η άλλη χώρα με τα συναφή. Είναι έτσι ή κάνω λάθος. Ευχαριστώ. Σταμάτησα. θα είμαι πολύ σύντομος. Τα θετικά μηνύματα που θέλουμε να δώσουμε στους Λετονούς είναι απλά. Δηλαδή, ε, την εποχή αυτή που υπάρχουν τόσο πολλά αρνητικά στοιχεία και πληροφορίες για διάφορες οικονομίες, η υποστήριξη 33% και 33% αναποφάσεις τη σημαίνουν στην ουσία μεγάλη υποστήριξη. Και η κεντρική μας τράπεζα και η κυβέρνηση δεν έχουν αρχίσει καμία καμπάνια, απλώς απαντάμε σε ερωτήσεις και απορίες. Όλοι αρχίζουν σιγά σιγά να καταλαβαίνουν ότι η Λετωνία θα μπει στην Ευρωζώνη και ενδιαφέρονται να έχουν τις πληροφορίες αυτές. Και εμείς θα τις χορηγήσουμε μέχρι το καλοκαίρι. Νομίζω ότι η πλειοψηφία θα υποστηρίζει το ευρώ, όπως έγινε και για την ένταξή μας στην Ένωση το 2003. Αντίθετα από μερικές χώρες που βρίσκονται ήδη στην Ευρωζώνη, σε εμά υπάρχει μεγάλη υποστήριξη και αυξάνεται για την ένταξη στην Ευρωζώνη. Το να μπούμε ή να μην μπούμε θα το, κρίνουμε, θα το κρίνει, πρέπει να το κρίνει κανείς σε σύγκριση και με ανοιχτές και κλειστές οικονομίες μεγάλες και μικρές. Εμείς είμαστε μία μικρή ανοιχτή οικονομία. Το 8 και το 9 τιμωρηθήκαμε γιατί ήμασταν απομονωμένοι, δεν είχαμε σταθερή ισοτιμία και μας επιτέθηκαν όλοι και περίμεναν να πέσουμε. Αν ήμασταν σε μεγαλύτερο πλοίο όπως οι μικρές χώρες που μπήκαν στην Ευρωζώνη πριν από εμά, τότε νομίζω ότι οι κερδοσκοπικές επιθέσεις δεν θα είχαν πετύχει. Γιατί η Λετωνία θα ήταν τότε σε θέση, αν ήταν από το 8 στην Ευρωζώνη, να διευθετήσει τα του δημοσιονομικού της οίκου και η καταιγίδα θα ήταν πολύ μικρότερη αυτή που υποστήκαμε. Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία του γιατί η Λετωνία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωζώνη για να μην υφίσταται κερδοσκοπικές επιθέσεις κατά το νομίσματός της στο μέλλον. Και νομίζω ότι η ένταξη αυτή προετοιμάζεται πολύ θετικά. Μάλιστα. Τώρα περνάμε στους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίζω και τους ε, προσκεκλημένους μας. Ε, το Κοινοβούλιο βεβαίως ε, υπερψήφισε την ένταξή σας, αλλά η πλειοψηφία είναι ισχνή, το είπαν ε, και άλλοι ομιλητές ε, ε, εντός της Λετωνίας και το ερώτημα είναι εφόσον έχει και το ευρώ μια δύσκολη κατάσταση γιατί βιάζεστε να ενταχθείτε υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για αυτή τη βιασύνη ναι είναι δύσκολο να, να απαντήσω πότε θα λυθούν τα ζητήματα της Ευρωζώνης. μπορεί να περιμένουμε χρόνια. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι πως πέρσι πολλές από τις χώρες ε, της Ευρωζώνης ε, έδωσαν προσοχή στην ε, εφαρμογή των μέτρων λιτότητας και μεταρρυθμίσεων και υπήρξε κάποια μεταστροφή καλοκαίρι προς φθινόπορο και έκτοτε οι αγορές δίνουν καλύτερα μηνύματα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε βεβαίως πως ε, θα απαιτηθούν ε, πολλά χρόνια προσπαθειών από πολλές χώρες και από ολόκληρη την Ευρωζώνη. Αλλά το να περιμένουμε χρόνια και να σπαταλάμε χρόνο δεν είναι η καλύτερη λύση για μικρές και ανοιχτές οικονομίες. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες ε, να είμαστε εντός της Ευρωζώνης και να λύσουμε από κοινού αυτά τα προβλήματα. Συν το ότι ε, θα είναι και καλό για την οικονομία μας, ε, θα είναι θετικό στοιχείο. Για ζητήματα ανάπτυξης ε, οικονομίας σε μια κοινωνία είναι σημαντικό στοιχείο. Δεν θέλουμε να περιμένουμε κάποιο μαγικό έτος όταν δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Είναι δύσκολο να να το κρίνουμε και είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε και να λύσουμε μαζί αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα δεν θέλετε να επανέλθετε. Περνάμε στο Έλκ και στον Κρίστιαν Κάρνς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε. Πως ε, είχε, όταν είχε μεγάλη ανάπτυξη η Λετωνία αυτή χρηματοδοτήθηκε κυρίως από χρέος και τη φούσκα των ακινήτων και όταν ε, σταμάτησε το Βλέδι όλα αυτά κατέρευσαν. Μπορείτε να μας περιγράψετε την διαφορά στην τωρινή ανάπτυξη σε σύγκριση με την ανάπτυξη προκρίσης. Ποια είναι η ουσιαστική διαφορά και γιατί θεωρείτε πως αυτή τη φορά είναι βιώσιμη αυτή η ανάπτυξη. Πράγματι, αυτή είναι η αλήθεια. Η ανάπτυξη του 2004-2007 βασιζόταν στον τομέα των κατασκευών και στο λιανεμπόριο, δανεισμός, εισαγωγές και υπερθέρμανση της οικονομίας. Αυτή τη φορά είναι τελείως διαφορετικά. Η ανάπτυξη βασίζεται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, βαριά βιομηχανία, μηχανολογικός εξοπλισμός, υφάσματα, μεταφορές, ε, τηλεπικοινωνίες. Γι' αυτό θεωρούμε πως είναι βιώσιμη. Βλέπουμε κάποιες αυξήσεις των μισθών και αυτή τη φορά δεν είναι 20-30% όπως ήταν τότε. Είναι μεταξύ 3 και 4% και κάποιες φορές 5% και συνδέεται με μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας. Μάλιστα. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Ωραία. Ελκ Βέρνερ Λάγγεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αντίθεση με τον Έλληνα κομμονιστή συνάδελφο, εγώ χαίρομαι για την πορεία που ακολούθησε η Λετωνία για το ότι είχατε επιτυχίες επί σειρά ετών και η Ελλάδα νομίζω πρέπει να παραδειγματιστεί από τη Λετωνία και όχι το, το αντίστροφο. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την πορεία που ακολουθείτε και βεβαίως γνωρίζουμε και τον Πρωθυπουργό που ήταν ε, επί σειρά ετών Ευρωβουλευτής, ξέρει πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Γι' αυτό ως Γερμανός Ευρωβουλευτής χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι θα έχουμε ένα νέο μέλος σε μια φάση ε, στην οποία δεν μιλάμε για την κρίση του ευρώ ως νομίσματος, αλλά για την έλλειψη ανταγωνιστικότητας και την μη ε, ορθή εκτέλεση των προπολογισμών κάποιων καρτών μελών. Ανεξαρτήτως τώρα των επένων, έχω τρία ερωτήματα. Τι γίνεται με την ενεργειακή εξάρτηση της ε, Λετωνίας ε, από όταν ε, έκλεισαν τα πυρηνικά εργοστάσια. Δεύτερον, τι κάνετε με τα προβλήματα των μειονοτήτων. Και τρίτον, πώς είναι προετοιμασμένος ο τραπεζικός τομέας για την τεχνική ε, μεταστροφή για την αλλαγή του νομίσματος. Θα τα καταφέρετε. Για τις δε θέλω να αναφέρω τον αριθμό των ε, απάτριδων ε, πρώην υπηκών της Έσουσουδού. Τι θεωρείτε, τι επίδραση θεωρείτε πως θα έχει αυτό μακροπρόθεσμα. I will uh, ξεκινήσω με την ενέργεια που είναι σημαντική για όλες τις βαλτικές χώρες. Ε, εξακολουθούμε να εξαρτώμεθα από τις προμήθειες αερίου από μία εταιρεία στη Ρωσία, αλλά αν δούμε τι γινόταν πριν από λίγα χρόνια, είχαμε προβλέψει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση και ανάγκες ενέργειας. Τώρα λοιπόν που ξεπεράσαμε το επίπεδο προκρίσης ε, σε κάποιες βιομηχανίες και τις κατασκευές χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια. Άρα γινόμαστε όλο και πιο αποτελεσματικοί στη χρήση της ενέργειας. Ε, αλλά ε, η λύση είναι δίκτυα, σύνδεση με τη σκανδιναβική αγορά και με την Πολωνία. Κοιτάμε διάφορες ανανεώσιμες. Στο επίπεδο των ανανεώσιμων είμαστε πολύ ψηλά. Δεύτερη μετά τη Σουηδία 40% αλλά πράγματι το πρώτο θέμα είναι η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Χάρη στα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, κάνουμε αυτή τη χρήση, όπως είπα, για τη θέρμανση των σπιτιών και την εξοικονόμηση της ενέργειας, αλλά θα είναι μια συνολικότερη βαλτική λύση. Είμαστε ήδη ανοιχτή και θα ανοίξει και άλλο η αγορά της ενέργειας στις βαλτικές χώρες και όπως σας είπα θα είναι συνολικά βαλτική η λύση και η συνεργασία. δεν ξέρω ε, το τι θα γίνει με τα, τα πυρνικά εργοστάσια. Τώρα για τις μειονότητες δεν είναι αυτό το, το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Αν δείτε την ε, πληθυσμιακή σύνδεση της και τα δικαιώματα δεν νομίζω πως υπάρχουν εντάσεις ε, για τέτοια πράγματα. Καμιά φορά κάποιες μεγάλες γειτονικές χώρες θέλουν να επηρεάσουν την κατάσταση στη Λετωνία, αλλά σε σύγκριση με άλλες ε, νομίζω περιοχές στην Ευρώπη, νομίζω πως έχουμε θετικές εξελίξεις στη Λετωνία. Να μιλήσω για τον τραπεζικό τομέα. Θα έλεγα πως 75% ε, των τραπεζών είναι σε ξένα χέρια, κυρίως ε, σκανδιναβικής ιδιοκτησίας. Οι τράπεζες παρέμειναν σταθερές ε, καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, ανακεφαλαιοποιήθηκαν. Αυτή τη στιγμή το, τα βασικά κύρια ίδια κεφάλαια είναι γύρω στο 50% και η ρυθμιστική αρχή εξετάζει τις πιο επισφαλείς καταθέσεις ε, μη ε, μονίμων κατοίκων δηλαδή. Οι τράπεζες είναι επικερδείς ε, και έχουν ρευστότητα. Οπότε θα έλεγα πως είναι καλά προετοιμασμένες για την μετάβαση στο ευρώ. Εάν λοιπόν ε, λάβουμε την πρόσκληση για ένταξη στο ευρώ θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τη μετάβαση για τα πρακτικά της μετάβασης Ευχαριστώ. Περνάμε στους σοσιαλδημοκράτες και τον κύριο Πάνταρ. Τους, ε, λόγω σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους γείτονές μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που έχετε κάνει. Εγώ ήμουν Υπουργός Οικονομικών της Εστονίας το 2008 και γνωρίζω τι αποφάσεις έπρεπε να λάβετε και πόσο δύσκολο ήταν θα μπορούσαμε να γράψουμε ολόκληρο βιβλίο για το πώς ε, μαζί μπορέσαμε να ε, νικήσουμε τον σκεπτικισμό που κρατούσε στο Δουνουτού και να πώς αποδείξαμε πως υπάρχει άλλος τρόπος. Συγχαρητήρια λοιπόν και ταυτόχρονα πολλά ευχαριστώ για τη διαδικασία αυτή. Πολλά ερωτήματα έχουν ήδη απαντηθεί και γι' αυτό ίσως θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που ήδη αναφέρθηκε, ότι δηλαδή έγινε πολλή κουβέντα για το ότι ο αριθμός των καταθέσεων από μη από πολίτες ε, ξένους, όπως Κύπροι ας πούμε, που έχουν πολλές καταθέσεις στη Λετωνία, ε, έχουν αυξηθεί. Τι μπορεί να κάνει η Λετωνία για να βλύνει τους κινδύνους που συνδέονται με αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ. Την περασμένη εβδομάδα μαζί με τον επόπτη Ήδη προβλέψαμε μια αναπάντηση και προσπαθήσαμε να εξαλείψουμε τον μύθο σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα της Λετωνίας, το οποίο ελκύει ε, τις καταθέσεις. Δεν είναι αυτό το κατάλληλό μας ε, μοντέλο, το πρότυπό μας, να ζούμε δηλαδή με βάση τις καταθέσεις των ε, αλλοδαπών. Λόγω τώρα, μάλλον για ιστορικούς λόγους, είχαμε ψηλά επίπεδα ξένων καταθέσεων ανάμεσα στο 40% και το 50% ανέκαθεν. Κατά τη διάρκεια της κρίσης μειώθηκαν και τώρα που βελτιώνεται η κατάσταση ανέβηκαν οι ξένες επενδύσεις στο 48%. Θα ήθελα να πω ότι το να συγκρίνουμε, το πιο σημαντικό, μάλλον όταν συγκρίνουμε, είναι να δούμε πως το μέγεθος τραπεζικού μας συστήματος είναι 132% σε σχέση με το ΑΕΠ και σε σχέση με το 300 περίπου τις 100 που είναι σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και με τους φίλους μας Κύπρους το, η αντιστοιχεία ανέρχεται στο 700% του ΑΕΠ τα κυπριακά χρήματα στη Λετωνία είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια περίπου. Οπότε έτσι έχετε μια εικόνα για τα μεγέθη για τα οποία μιλάμε. Πρόσφατα ελέγξαμε αν υπήρξαν ροές από την Κύπρο προς την Λετωνία, αλλά αυτές είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Οπότε μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η Λετωνία ποτέ δεν προσπάθησε να αποτελέσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις, ε, ξένες μάλλον καταθέσεις, αλλά ε, σαφώς αναφέρεται στο τελευταία έκθεση για, τους, ε, για, για τις χρηματικές συναλλαγές και ε, την έχουμε στείλει την έκθεση αυτή ώστε να γνωρίσουν καλύτερα την κατάσταση της Λετωνίας, ότι δηλαδή εμείς πληρούμε όλες τις συστάσεις, έχουμε, δεν είμαστε στον κατάλογο των χωρών που δεν πληρούν τις ε, συστάσεις. Σας ευχαριστώ. Τώρα, ο Γκέι Μίτσελ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους μας. Όταν ακούω την ιστορία της Λετωνίας μου θυμίζει το σχόλιο που λέει όλα ωραία ε, και καλά, λειτουργούν στην πράξη, αλλά... Ναι, ναι τι γίνεται με την ε, ε, ε, χώρα. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι πραγματικά είναι αξιοσημείωτα τα όσα έχετε καταφέρει, όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και ο λαός της Λετωνίας και αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Τα επιτεύγματα είναι ε, πολύ σπουδαία. Επίσης ε, συμφωνώ με τα σχόλια ότι η Ιρλανδία, ε, ότι η Λετωνία όπως και η Ιρλανδία προσπαθεί να βρει εσωτερικές λύσεις δικές της και όχι να αντιγράψει λύσεις που έχουν εφεύρει μεγαλύτερες χώρες. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Η Λετωνία και η Λιθουανία για λίγο δεν ε, μπορούν ακόμα να μπουν στο ευρώ. Αν δεν μπείτε, θα χάσετε το τρένο της ανάκαμψης. Αυτό το εξηγείτε αρκετά στο λαό της Λετωνίας. Και έπειτα η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας ε, και διαπιστώνω πως όλα αυτά έχουν αλλάξει μέσω νομοθεσίας αλλά θα μπορούσε να ξαναλλάξει σχετική νομοθεσία ή πια αυτά είναι απόλυτα καθορισμένα. Στη χώρα μου ας πούμε αυτά έχουν εγγραφεί στο Σύνταγμα. Έχει γίνει κάτι παρόμοιο και στη Λετωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις πολύ σημαντικές ερωτήσεις σας. Θα έλεγα ότι κανείς αυτή την αίθουσα θα πρέπει να ανησυχεί για την εξαρτησία της κεντρικής μας τράπεζας. Η κεντρική τράπεζα της Λετωνίας είναι μια από τις πιο ανεξάρτητες σύμφωνα με την έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ε, η άλλη πιο ανεξάρτητη είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι αλλαγές που έγιναν πρόσφατα στόχο είχαν να εναρμονίσουν τη διατύπωση που περιλαμβάνεται στο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή δεν ε, αποδυναμώνεται η ανεξαρτησία της Κεντρικής μας Τράπεζας. Για τη δεύτερη ερώτηση, όπως αναφέρθηκε ήδη τώρα στο ο Υπουργός, δεν βιαζόμαστε να μπούμε στην ε, Ευρωζώνη. Δεν είμαστε απελπισμένοι είναι μια φυσιολογική διαδικασία ε, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή ε, η Λετωνία από το 2005 λέει ότι θα μπει στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και σύμφωνα με το καταστατικό και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες από τη στιγμή που μια χώρα είναι έτοιμη πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Και όπως εξήγησε ο Υπουργός μας, δεν βλέπουμε για ποιο λόγο πρέπει να περιμένουμε, να μένουμε εκτός αφού θέλουμε να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία, θέλουμε να είμαστε κοντά και να οικοδομούμε την Ευρώπη όλοι μαζί. Μάλιστα. Προχωρούμε. Σαμπεν Κούτας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ και εγώ τη Λετωνία για τις προσπάθειες που έχει κάνει για να ενταχθεί στην Ευρωζώνη. Υπάρχουν ακόμη βέβαια μερικά προβλήματα, αλλά είμαι βέβαιος ότι η Λετωνία θα καταφέρει να γίνει το υπόδειγμα των βαλτικών χωρών για την ένταξη στην Ευρωζώνη. Επειδή εγώ είμαι Ρουμάνος, αντιμετωπίζουμε παρόμοια προβλήματα, όχι τα ίδια, αλλά παρόμοια και με ενδιαφέρει πολύ η εμπειρία σας και το πώς αντιμετωπίσατε το πρόβλημα. Ερωτώ λοιπόν, Ποια είναι η κυριότερη σύσταση που έχετε να κάνετε για μια χώρα που και αυτή θέλει να ενταχθεί και τι θα είχατε κάνει καλύτερα, τι λάθη θα είχατε αποφύγει. Γιατί εμείς στη Ρουμανία αντιμετωπίζουμε τις ίδιες αμφιβολίες του πληθυσμού για την ένταξη στην Ευρωζώνη όχι μόνο λόγω των προβλημάτων της και γι' αυτό ερωτώ τι συστήνεται σε μια χώρα που θέλει και αυτή να ενταχθεί. Μα υπάρχουν ήδη βιβλία για αυτά και για την περίπτωσή μας από κάποιο Σουηδό νομίζω γράφτηκε. Τα προβλήματα που είχαμε πρόσφατα ήταν τεράστια και γι' αυτό θελήσαμε να δούμε τι είναι αυτό που έπρεπε κατά προτεραιότητα να γίνει. Αυτό που χρειάζεται είναι η λήψη τολμηρών αποφάσεων για να βγει κανείς από την κρίση. Και καταλάβαμε ότι ως μικρή χώρα έπρεπε να είμαστε αποτελεσματικοί. Κύριο, θέμα είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. και η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική, η επικοινωνία. Πρέπει οι πολιτικοί να συνεννοηθούν. Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπα και πριν, ο κοινωνικός διάλογος. Πάρα πολύ σημαντικό. Αν τα συνδικάτα και οι επιχειρηματίες καταλάβουν ότι μόνο μαζί θα λυθούν τα προβλήματα, είναι πολύ σημαντικό και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις Παντού στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, χρειάζονται. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει ανταγωνιστικότητα, μειώνεται η ανταγωνιστικότητά της. Και εδώ το θέμα είναι πώς θα πείσουμε την κοινωνία. Είναι θέμα επικοινωνίας. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει καλή επικοινωνία σε καιρούς κρίσης. Μας έχουν δώσει συμβουλές από το Δουνουτού, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από άλλες χώρες. Τα συνδυάσαμε όλα αυτά και θελήσαμε να προοδεύσουμε. Κυρίως μας είπαν να επιδείξετε τόλμη και να μην σπαταλήσετε χρόνο. Καταφέραμε να επιδείξουμε ευελιξία και όλη η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη ευελιξία. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω να χρησιμοποιήσετε τη λογική σας και να μην ακούτε τους νομπελίστες που λένε ότι η α ή η β χώρα σε έξι μήνες ή τρία χρόνια θα πτωχεύσει. Εδώ χρειάζεται νέου είδους σκέψη και υπάρχει, υπάρχει. Um, πολύ ωραία. Λοιπόν, για το ΕΛΚ τώρα. Κορίν Βόρτμαν Κόλ, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ, κύριε Διοικητά, μαζί με τους συναδέλφους θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ για αυτά τα οποία επιτύχατε για τον λαό της Λετωνίας και βεβαίως αναγνωρίζουμε πως η κατάσταση είναι ακόμα πολύ δύσκολη για πολλούς ανθρώπους στην χώρα σας, αλλά είναι εκπληκτικό το ότι έχετε επιτύχει μια πορεία προς βιώσιμη ανάπτυξη και δεν είναι αποφασιστικό μόνο, μόνο τα στοιχεία του προϋπολογισμού, αλλά είχατε και το θάρρος να κάνετε μεταρρυθμίσεις που δεν είναι εύκολες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εδρεωμένα συμφέροντα αλλά το κάνατε αυτό και με κοινωνικό διάλογο. Αυτό νομίζω είναι βασικός παράγοντας της επιτυχίας. Και βλέπουμε τι γίνεται και στην Ιρλανδία όπου αποδίδει και αυτό νομίζω έχει μεγάλη σημασία για να έχουν στήριξη οι πολιτικές σας και να έχουν θετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα τώρα με το ερώτημά μου να ασχοληθώ με τον τραπεζικό τομέα και το πώς πηγαίνει αυτό. Στην προηγούμενη εβδομάδα ήταν στην Επιτροπή μας ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής, ο διοικητής Ευρωπαϊκής και ο κύριος Δράγκη, ο οποίος μας είπε πως το μεγάλο πρόβλημα είναι πως η ρευστότητα δεν περνάει από τις τράπεζες στην πραγματική οικονομία. Δεν είστε ακόμα εντός της Ευρωζώνης, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι πως μιλήσατε για την κερδοφορία, τη ρευστότητα του τραπεζικού τομέα σας, αλλά α, τα λεφτά διοχετεύονται στις επιχειρήσεις στην πραγματική οικονομία. Σας στηρίζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα άλλα πιστοτικά ιδρύματα για να ξεπεράσει τα προβλήματα αυτά. Χαίρομαι για την ερώτηση αυτή, γιατί αυτή η ερώτηση είναι πραγματικά το κλειδί της ε, συζήτησης για το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα γιατί μεγάλο μέρος της ρευστότητα ακόμα δεν ε, διοχετεύεται στην πραγματική οικονομία γιατί δεν έχουν υπάρξει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, γιατί υπάρχουν φορολογικά προβλήματα, γιατί οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες περιμένουν το εάν θα έχουμε μείωση των δαπανών ή αύξηση της φορολογίας. Και αν ακολουθήσουμε την αύξηση της φορολογίας, γιατί εγώ ως τράπεζα να δανείσω σε μια επιχείρηση αν αύριο αυτή δεν θα είναι κερδοφόρα και ε, ίσως φαλυρίσει. Πριν λοιπόν τακτοποιήσουμε τα του φορολογικού οίκου μας ε, και μας να μας πιστέψουν οι τράπεζες, οι τράπεζες θα κρατάνε τη ρευστότητα και δεν θα δανείζουν στις επιχειρήσεις. Για τη Λετωνία τώρα βλέπουμε πως υπάρχει μια αλλαγή στην σκέψη, στην οτροπία. Βλέπουμε πως τα δάνεια στα νοικοκυριά ε, είναι στάσιμα και μειώνονται κιόλας γιατί υπάρχει ακόμα απομόχλευση από τα πολύ υψηλά επίπεδα της κρίσης αλλά βλέπουμε πως ο τομέας των επιχειρήσεων ανακάμπτει ε, διοχετεύονται λεφτά εκεί πέρα και επανέρχεται ο δανεισμός. θέλετε να επανέλθετε για το δεύτερο τμήμα της ερώτησης για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων λειτουργεί και από άλλα επίσης ε, ιδρύματα όσον αφορά την παροχή δανείων και τα λοιπά. Ναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά κονδύλια είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του οικονομικού μας συστήματος και είναι, πάει χέρι-χέρι με την υγεία της οικονομίας. Εάν οι τράπεζες είναι διατεθειμένες να δώσουν ε, ένα αρχικό κεφάλαιο ή μια προκαταβολή ή μια αρχική χρηματοδότηση, οπωσδήποτε και η... τα χρήματα αυτά βέβαια ευκολότερα διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία. Ευχαριστώ και η τελευταία μας ερώτηση από τον Βολφ Κλίντς, από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα ερώτημα στον ε, διοικητή και ένα στον κύριο Υπουργό. Τι άποψη έχετε για αυτό το οποίο λέγεται για την Ευρωζώνη για κοινή έκδοση ομολόγων. Είστε κατά. Και θα φέρετε ένα φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών όπως έχουν κάνει 12 χώρες και τι σκοπεύετε να κάνετε για να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με κάποιες άλλες χώρες της ε, περιφέρειας. Η Κομισιόν παραδείγματο χάρη σκοπεύει να στείλει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να αποστείλετε εσείς ειδικά νομίζω εμπειρογνώμονες. Ναι. Η Λετωνία είναι ε, νομίζω έτοιμη να ενταχθεί στην ομάδα των χωρών εκείνων που θα εφαρμόσουν τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ε, και πάλι όμως η Ευρώπη πρέπει να προσέξει να μην χάσει σε παγκόσμιο πλαίσιο ανταγωνιστικότητα. Είμαστε έτοιμοι, όπως είπα, να προχωρήσουμε και εμείς. Αυτό το οποίο έχουμε είναι το λεγόμενο τέλος το χρηματοπιστωτικό, το οποίο το διπλασιάσαμε. Οπότε υπάρχει ήδη κάποιο είδους ε, φόρος τέτοιος. Το εάν θα εισαχθεί ο συγκεκριμένος αυτός φόρος εξαρτάται και με το τι θα κάνουμε με το αντίστοιχο τέλος για να μην μειωθεί η ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού μας τομέα σε σύγκριση με άλλες χώρες, αλλά είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα και είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσον, ε, εάν γίνει σωστή διαχείριση θα έλεγα. Το ερώτημα για τα ευρωομόλογα έχει νομίζω απαντηθεί. Όσοι ασχολούνται με οικονομικά ζητήματα γνωρίζουν πως ε, τα ευρωομόλογα θα είναι ένα μέσο επιδότησης και όλοι μπορούν εύκολα να υπολογίσουν ε, πόσα χρήματα θα πρέπει να πληρώσει κάθε χώρα στην περίπτωση των ευρωομολόγων. Οπωσδήποτε εμεί θεωρούμε πως ε, τα ευρωομόλογα θα είναι αντικίνητρο για τις χώρες για να κάνουν ε, αυτά που χρειάζονται για να τακτοποιήσουν τα οικονομικά τους και άρα μακροπρόθεσμα θα βλάψουν την ε, δημοσιονομική σταθερότητα. Κάτι ακόμα είναι ε, που δεν απαντήθηκε. Η Κομισιόν σας ζήτησε να βοηθήσετε ε, άλλες ε, χώρες της περιφέρειας να μοιραστείτε την εμπειρία σας. Σας ζήτησε να πάτε στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία κτλ. για να μοιραστείτε την εμπειρία σας. Ναι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν ήδη εμπλακεί στην ομάδα της Κομισιόν που εδρεύει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Ναι. Μάλιστα. Τελειώνει λοιπόν εδώ πέρα η ανταλλαγή απόψεων με τους ε, προσκεκλημένους μας από την Λετωνία. Σας ευχαριστώ όλους. Περνάμε τώρα στις ανακοινώσεις. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 2-3 λεπτών μέχρι να μοιραστούν τα σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε σε λίγο.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 Um, Τα άσχημα νέα είναι ότι έχω να κάνω κάποιες ανακοινώσεις του Προέδρου. Θα προσπαθήσω να το κάνω όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τώρα για την AIFM deal δεύτερο επίπεδο. Η προθεσμία που έχει θεσπίσει η γραμματεία μέχρι ότου δηλαδή μπορείτε να εκφράσετε αντιρρήσεις για κατεξοδότηση πράξης το ζητήσαμε να είναι 27 Ιανουαρίου. Δεν έχει υποβληθεί τίποτα. Άρα λοιπόν το άρθρο 27α του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να κατατεθεί αντίρρηση, αλλά η Γραμματεία δεν γνωρίζει κάποια τέτοια πρόθεση ή πρόταση. Εάν δεν υπάρξει περαιτέρω ενέργεια, η προθεσμία για αντίρρηση εκπνέει για το Κοινοβούλιο στις 19 Μαρτίου. Ενημέρωση για τους συνεχιζόμενους τριμερείς διαλόγους. Έχουμε τρίτο τριμερή διάλογο που έγινε στις 20 Φεβρουαρίου. Ε, νέες διατάξεις συζητήθηκαν όπως η εξολόγηση ιδιοκτησίας, τα δίκτυα σε ξενονόμισμα, ε, καθώς και οι απαιτήσει για δεξιότητες ή πτυχία. Περαιτέρω διατριμερή διάλογο θα γίνει στι 19 Μαρτίου. Βέρνερ, εσύ με, μου κάνει να είμαι ποιο, για ποιο θέμα είναι. Ναι, πράξει κατά Η Κομισιόν μα είχε υποσχεθεί πω ε, η επόμενη πράξη κατά εξουσιοδότηση θα είχε υποβληθεί μέχρι τέλο ε, Ιανουαρίου για την ε, ΕΜΕΑ. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι τέλος Φεβρουαρίου πρέπει να το συζητήσουμε. Υποτίθεται Στρασβούργο. Παρακαλώ λοιπόν να απευθυνθείτε να γράψετε μια επιστολή στην Κομισιόν. Okay, we, we take note of that. Um, Ωραία, το σημειώνουμε. Στρεφόμαστε στους τριμερείς διαλόγους και στην οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις έγινε τριμερείς διάλογος 19 Φεβρουαρίου πέρα από τη συζήτηση της ενημέρωσης που μας έδωσε η τεχνική ομάδα για θέματα όπως ε, προληπτικά φίλτρα, ορισμός ε, των ε, όρων περί επενδύσεων. Ήταν η σειρά του Συμβουλίου να επανέλθει για να δούμε αν χρειάζεται να, να θεωρήσουμε τις συμβαστικές που είχαν εξευρεθεί από την Κυπριακή Προεδρία. Τα θέματα που θέλουν να ξανανοίξουν είναι οι αμοιβέ, η μακροπροληπτική ευελιξία, επιπλέον κεφαλαία και φραγμή για τις ε, χώριες σημαντικές ε, ε, τράπεζες και ε, από την άποψη του Κοινοβουλίου πρέπει να βρεθεί ικανοποιητική λύση για τα θέματα αναχώρας έκθεσης ε, όσον αφορά τα κέρδη, τους φόρους και τις επιδοτήσεις στις μεμονωμένες χώρες. Η διαπραγματευτική μας ομάδα ελπίζει ότι τα τελευταία κρεμή ζητήματα θα ρυθμιστούν στην επόμενο τριμερή διάλογο στις 27 Φεβρουαρίου, δηλαδή αύριο. Ακόμα και αν κάτι τέτοιο δεν ε, συμβεί, μετά από 10 μήνες διαπραγματεύσεων και τρεις προεδρίες είναι και πλέον η ώρα να προχωρήσουμε στην Ολομέλεια. Έβδομος δε τριμερής διάλογος έγινε στις 27 ε, Ιανουαρίου για το θέμα της EBA ε, και επόμενη συνάντηση προβλέπεται σήμερα το απόγευμα με στόχο να εξεταστούν τα εκκρεμή πολιτικά ζητήματα στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης, περισσότεροι νέοι κανόνες, νέα πράγματα πρέπει να ανακοινώσω στη συνάντηση στις 24 Ιανουαρίου. Οι συντονιστές συμφώνησαν για την ανάθεση νέων διαδικασιών. Το FTT πάει στους σοσιαλιστές, είναι η πρόταση για την ουσία της αυξημένης συνεργασίας, της ενισχυμένης συνεργασίας ο κανονισμός ε, για τη μεταφορά επιβατών οδικός και σιδηροδρομικός ανατίθεται στο ΕΛΚ, οι κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 93 επίσης στο ΕΛΚ, το πρόγραμμα της Ένωσης στον τομέα της έκθεσης και ελέγχου των οικονομικών στο ΕΛΚ, οι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ECR, ετήσια έκθεση 2012 της ΕΚΤ στους σοσιαλιστές, ετήσια έκθεση περιενταγωνισμού 2012 στην Άλντε, γνωμοδότηση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στους Σοσιαλιστές, προϋπολογισμοί και γνωμοδοτήσεις για τον προϋπολογισμό του 2014 στους Πρασίνους, ε, χρηματιστήρια γνωμοδότηση είναι αυτή για την ΑΛΔΕ. στις 5 Φεβρουαρίου υιοθετείται από την Λετωνία το ευρώ στο ΕΛΚ και νομοθετικός έλεγχος, οι νομοθετικές αρμοδιότητες για τις κατεξοδότησες πράξεις από και των μελών ε, ε, γίνεται από την Προεδρία. Αυτά λοιπόν, να βρούμε τώρα και τις ε, ψηφοφορίες. Okay, and the first vote is the Agenda point five. We'll just have the secretariat shuffle. Πρώτο σημείο ε, η, το 25 κοινό σύστημα ΦΠΑ όσον αφορά τα vouchers. Λοιπόν, συμβαστική α, ποιοι είναι υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ε, ε, το 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Γ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, εκτιμώντας 1, τροπολογία 9, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική δέλτα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε unblock νομίζω για τις τροπολογίες 12 μέχρι και 16. Όχι δεν μπορούμε. Ωραία. 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, απορρίπτεται με συγχωρείτε ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε. Συγχρεμία. Λοιπόν. Τέλος της ψηφοφορίας. 40 υπέρ και μια αποχή. Και τώρα ψηφίζουμε για το νομοθετικό ψήφισμα. Τέσσερα ακόμα κουμπάκια. Ευχαριστώ. 43 υπέρ. Κανείς κατά. Καμιά αποχή. Συγχαρητήρια στο συντάκτη. Right, uh, we've Ωραία. Τελειώσαμε με αυτό. Υπάρχει πρόβλημα. Ναι, να σας ρωτήσω κυρία Πρόεδρε πρέπει να προσθεθεί άλλη μια ψήφος ε, στην ε, τελική ε, ψηφοφορία γιατί δεν λειτουργούσε η κάρτα μου για το πρώτο έτσι στο δεύτερη φορά ψήφισα την πρώτη δεν μπορούσα μάλιστα οπότε είναι 44 ωραία μάλιστα θα, θα αλλάξουμε το αποτέλεσμα 44 υπέρ κανείς κατά Α, στην πρώτη ψηφοφορία. Στην πρώτη. Εντάξει. Περνάμε τώρα στις ε, επαρκείς ε, ασφαλείς και βιώσιμες ε, συντάξεις. Έχουμε προφορική τροπολογία του εισηγητή επί του τίτλου 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή Οπότε καταπίπτει η τροπολογία 1. Πάμε στην παράγραφο 1 του αρχικού κειμένου υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 2 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω. Θα το επαληθεύσουμε. Το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 2. Άρχεται ψηφοφορία. Τώρα είναι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Κάποιος από το ΕΛΚ πρέπει να βγάλει την κάρτα. Ευχαριστώ. Πέρας. 18 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβαστική α υπέρ, κατά αποχές δεκτή προφορική τροπολογία στην παράγραφο 2α θα την ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές δεκτή τώρα τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε 19 Ψήφισαν ναι. όλοι, πέρας, ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές να την επαληθεύσουμε και αυτήν. Ψήφισαν όλοι. Δύο ακόμη μπορούν να ψηφίσουν. Ήταν ένας παραπάνω από το ΕΛΚ, αλλά είναι 24 με 16, οπότε δεν κάνει διαφορά, γίνεται δεκτή. Αλλά υπάρχει ένας παραπάνω από το ΕΛΚ πάλι. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή προφορική τροπολογία στον τίτλο 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή οπότε περνάμε στην παράγραφο 7 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική γάμα υπέρ κατά αποχές δεκτή 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές δεκτή 43 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε 43 Άλλη μία έχουμε να προσθέσουμε. Κάποιος δεν έχει κάρτα. Πέρας της ψηφοφορίας και γίνεται δεκτή. 26 με 18. 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική ε σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική σίγμα τάφα συμπεριλαμβάνει και προφορική τροπολογία του Όλε Λούντβιξεν δεχόμαστε την προφορική τροπολογία ναι υπέρ Να ψηφίσουμε την προφορική λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Εποχές δεκτή. Οπότε δεκτή η προφορική τροπολογία. Για να μην υπάρχουν λοιπόν αμφιβολίες. Θα δούμε τώρα όλοι μαζί την συμβαστική. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική ζήτα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική ήττα σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή. 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική θήτα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική γιώτα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Γιώτα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία του εισηγητή παράγραφος 17 υπέρ κατά, κατά αποχές δεκτή. 91 όχι. 91 καταπίπτει. Παράγραφος 18. Συμβιβαστική για τα β' υπέρ κατά αποχές δεκτή. 94 υπέρ κατά αποχές δεκτή να την επαληθεύσω την 94 συν ε, μία της περβάμψης ψήφισαν όλοι ωραία πέρας 26 υπέρ 19 κατά δεκτή λοιπόν προφορική τροπολογία στην παράγραφο 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 96 λοιπόν υπέρ κατά αποχές δεκτή 97 υπέρ κατά αποχές δεκτή 98 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική M υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική N υπέρ κατά αποχές δεκτή 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία του Τόμας Μαν στην παράγραφο 21. Είμαστε υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 106 καταπίπτει. Παράγραφος 22 συμβαστική όμκρον υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προφορική του εισηγητή στον τίτλο 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα στην παράγραφο 23, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική π υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία στην παράγραφο 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα στην 27 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο λοιπόν υπέρ κατά αποχές δεκτό παράγραφος 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 117 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως έγινε δεκτή θα την επαληθεύσουμε 117 συν υπερβάς είναι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ τώρα ένας παραπάνω από το ΕΛΚ ευχαριστώ πέρας απορρίπτεται γιατί και με την υπερβάς ακόμα είναι 22 υπέρ 23 κατά οπότε απορρίπτεται οπότε το αρχικό κείμενο της παραγράφου 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 118 υπέρ κατά αποχές δεκτή 119 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτή 120 υπέρ κατά αποχές δεκτή 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 122 δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε αλλά το αρχικό κείμενο άρα υπέρ κατά αποχές δεκτή 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό 124 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές δεκτή 127 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε 127 ψήφισαν όλοι δεκτή 26 με 19 προφορική τροπολογία στην παράγραφο 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή παράγραφος 35 συμβαστική άρη υπέρ κατά αποχές δεκτή παράγραφος 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο στις 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο στις 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή 134 υπέρ κατά αποχές δεκτή 135 υπέρ κατά αποχές δεκτή ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία ε, και την περιβάση να προσθέσουμε υπέρ δύο ακόμα πρέπει να ψηφίσουν ένας ακόμα πέρας 42 υπέρ, μία κατά καμία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν. Τώρα περνάμε στο σημείο, στα σημεία 7, 8 και 9. Πρώτον, η απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών του Βερνάρδου Λάγκεν. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά, ποχές αποδεκτό. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 πως πως όχι. Τρία, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 έχει αποσυρθεί. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, πρώτο τμήμα, όχι. Επειδή έχει εγκριθεί η 11, το πρώτο τμήμα έχει καταπέσει. Λοιπόν, το δεύτερο τμήμα της 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14, υπέρ, κατά, αποχές. Ορίστε. Α, έχει καταπέσει, α, μάλιστα. Και η 15. Επομένως το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί ηλεκτρονικά Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Λίγη ψηφοφορία. 42 υπέρ. Μία αποχή. Εγκρίθηκε. Μήπως θέλεις να λάβεις το λόγο. Βερνάρδο, όχι. Βάρνερ. όχι. Ωραία, επόμενη ψηφοφορία. Μα δεν ήθελες το λόγο, εντάξει. Λοιπόν, απλώς κουνούσε στα χέρια σου. Λοιπόν, απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Παράγραφος 1, αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται, 3 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 είναι γλωσσική. Το αρχικό της παραγράφου 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα της 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το κείμενο στο σύνολό του ηλεκτρονικά. Μάλιστα, έλξη ψηφοφορία. 43 υπέρ, μία αποχή. Τελευταία ψηφοφορία για την αρχή ασφαλής και επαγγελματικών συντάξεων. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 Αρχικό της 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά Κατά. Ψήφισαν όλοι. Έληξε 44 υπέρ μία αποχή. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ερχόμαστε στο σημείο 10. Μεταρρύθμιση της διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα. Τομέα. Ιδίας πρωτοβουλίας. Σχετίζεται με την έκθεση Λικάνεν αν η Κομισιόν εγκαίρως πει τίποτα θα το λάβουμε υπόψη μας. Η συγκήτρια είναι η Αρλίν και θα της δώσω αμέσως και τον λόγο. Α, σας ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη χαρά με τους σκιώδεις θα ήθελα να καταλήξουμε σε μία φιλόδοξη εργασία γιατί σε σχέση σε σύγκριση με τις προτάσεις που έχουν ήδη γίνει. Δεν θα επισελθώ σε λεπτομέρειες στις προτάσεις της υψηλής ομάδας Λίκανεν, απλώς θα τονίσω τα βασικά. Ο στόχος βέβαια ήταν να, εξεταστούν, να εξεταστεί η διαρθρωτική μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα της Ένωσης για να ανταποκριθούμε στην κρίση και μετά από μικρές διαβουλεύσεις και πολλές έρευνες υπευλήθη μία πρόταση για εφαρμογή σε πανενωσιακό επίπεδο. Αλλά βέβαια αυτό είναι ένα κομμάτι μόνο του παζλ της τραπεζικής μεταρρυθμίσεως. Στα πλαίσια των υπολείπων μεταρρυθμίσεων και βέβαια και οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν αναλάβει μεταρρυθμίσεις. Θα ήθελα λοιπόν απλώς να επαναλάβω τα πέντε κύρια στοιχεία της πρότασης. Υποχρεωτικός διαχωρισμός λιανικών και επενδυτικών τραπεζών με κύρια ιδέα να γίνει υποχρεωτικός ο προτινόμενος αυτός διαχωρισμός εάν οι δραστηριότητες και στους δύο τομείς έχουν κάποια σημασία βέβαια ποσοτικά. Δεύτερη πρόταση, και άλλος διαχωρισμός σε σχέση με τα σχέδια και προγράμματα αναδιάρθρωσης και αναθέρμανσης, εάν χρειάζεται. Τρίτον, η χρησιμοποίηση των διασωστικών μηχανισμών με στόχο την απορρόφηση των απολειών των σημειών από άλλες τράπεζες τέσσερα τα δανειοδοτικά. Uh, και τέλος πέμπτον, αλλά και εξίσου σημαντικό, η ενδυνάμωση της διακυβέρνησης και του ελέγχου των τραπεζών μέσω καταλήλων μηχανισμών στα διοικητικά συμβούλια, καλύτερο σχεδιασμό της ανάληψης κινδύνου, αποζημιώσεων πληροφόρησης για την ανάληψη των κινδύνων και περισσότερες και ισχυρότερες κυρώσεις. Όπως θα γνωρίζετε, η ομάδα αυτή θεώρησε δύο δρόμους δυνατούς. Ο πρώτος, πρόσθετο μη διακινδυνευμένο κεφάλαιο για τα προγράμματα διάσωσης των τραπεζών με κύριο όργανο τη μεταρρύθμισή τους, αλλά καταλήξανε ότι ο μόνος τρόπος να επανέλθουμε στην εμπιστοσύνη του κοινού είναι οι φορολογούμενοι να μην χρηματοδοτούν πλέον αμέσως ή εμέσως τις διασώσεις των τραπεζών. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να μιλήσουμε σαν μια πρώτη αρχή τουλάχιστον και βλέπω, προσβλέπω εδώ στους σκιώδεις να αναρωτηθούμε γιατί χρειάζονται οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Γιατί. Εδώ και πέντε χρόνια από την αρχή της δημοσιονομικής κρίσης η οικονομία της Ένωσης δεν βρίσκεται σε αναθέρμανση και ακόμα υποφέρει από τις επιπτώσεις της κρίσης όπως τα μέτρα λιτότητας και την υψηλή ανεργία. Και όλα αυτά έχουν κοστίσει στις ενωσιακές κυβερνήσεις 1,3 τρισεκατομμύρια περίπου. Αυτά είναι τεράστιο ποσό των χρημάτων των φορολογουμένων και κανείς δεν τα καταλαβαίνει και όλα στα μέτρα αυτά. Φυσικά μερικά από αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται μέσω της νομοθεσίας για το κεφάλαιο που απαιτείται για τη λειτουργία των τραπεζών, αλλά παρόλα αυτά ακόμα χρειάζονται διασώσεις. Σας υπενθυμίζω ότι στις αρχές του έτους η Ολλανδία εθνικοποίησε την τέταρτη μεγαλύτερη της τράπεζα για να ανακεφαλαιοποιήσει Παρακαλώ, λέει, θα λέτε πολύ γρήγορα, λέει η πρόεδρο, και δεν προλαβαίνουν οι διερμηνεύτριε. Λοιπόν, αυτό κόστησε 3,7 δισεκατομμύρια στην Ολλανδική κυβέρνηση και έτσι αυξήθηκε το έλλειμμά της. Άρα την ίδια κατάσταση αντιμετωπίζουμε και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Και μαζί με αυτό υπάρχει η έλλειψη εμπιστοσύνης στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. Γιατί δεν προωθεί την ανάπτυξη. Το Δεκέμβριο η Κομισιόν δήλωσε ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα, δεν έχουμε βγει από την τραπεζική κρίση και υπάρχουν στατιστικά στοιχεία και από οργανώσεις καταναλωτών στη χώρα μου τουλάχιστον η ομάδα WITS που βαθμολογεί την ικανοποίηση των καταναλωτών από τις τράπεζες έδειξε πολύ άσχημα αποτελέσματα. 70% δεν θεωρούν ότι πήραν το μάθημα που έπρεπε οι τράπεζες, ενώ προηγουμένως ήταν 61% τον προηγούμενο χρόνο. 11% μόνο έχουν εμπιστοσύνη στις τράπεζες και μόνο 6% από εκείνους θεωρούν ότι η συμπεριφορά των τραπεζών ακολουθεί την δέουσα δεοντολογία. Θεωρούν δε ότι πρέπει οι τράπεζες που παραβιάζουν τη δεοντολογία αυτή πρέπει να κλείνουν. Όταν λοιπόν εξετάζουμε τους στόχους της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης του τραπεζικού συστήματος της Ένωσης πρέπει να έχουμε ορισμένα ελάχιστα που πρέπει να στοχεύουμε. Δηλαδή, βιώσιμο και σταθερό τραπεζικό σύστημα που να περιορίζει την ανάληψη κινδύνου, να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση δημοσίου χρήματος για την αντιμετώπιση ιδιωτικών ζημιών να περιοριστεί η ανάληψη κινδύνου από τις καταθέσεις του κόσμου εκ μέρους των τραπεζών και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των λεγόμενων τραπεζών που είναι υπερβολικά μεγάλες για να πτωχεύσουν. Στη Γαλλία υπάρχει Λουάντε σε παρασιόν εντερεκιουλασιόν des activités bancaires. Στη Γερμανία υπάρχει το Trend Banking Gesetz και στο Ηνωμένο Βασίλειο η έκθεση για τις τραπεζικές μεταρρυθμίσεις που επίκυνται. Αυτή είναι διαφορετική δρόμη για την αντιμετώπιση του ίδιου προβλήματος. Η έκθεση Λικάνεν και η συζήτησή της στον τύπο βασίστηκε ιδιαίτερα στο θέμα της συγκέντρωσης και του διαχωρισμού των τραπεζικών δραστηριοτήτων από τον λιανικό και τον επενδυτικό τομέα. Αλλά θα έπρεπε ίσως να σκεφτούμε τα πράγματα ευρύτερα. Η συζήτηση αυτή να μην αφορά μόνο την περιορισμό της ανάληψης κινδύνων και την πρόληψη κρίσεων. Γιατί νομίζω ότι η δουλειά μας εδώ θα ήταν να διατυπώσουμε ιδέες για τη δημιουργία ενό σταθερότερου τραπεζικού συστήματος. Τι θέλουμε να κάνουν οι τραπεζέ μας και επομένως ποιε δομές διασφαλίζουν το στόχο αυτό. Θέλουμε σταθερότερη βάση λειτουργία των τραπεζών, όχι απλώς βιωσιμότητα αλλά και απελευθέρωση των τραπεζικών δραστηριοτήτων από την κρατική βοήθεια ώστε να υπάρχει εγγύηση των καταθέσεων και η αποταμίευση να κινείται προς ε, αναπτυξιακούς στόχους, στηρίζοντας την πραγματική οικονομία. Πράγμα το οποίο θα συνέβαλε στην αύξηση της σταθερότητας όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίω. Το θέμα αυτό λοιπόν του διαχωρισμού των τραπεζικών δραστηριοτήτων θέτει τα εξή με τη σειρά του προβλήματα. Πρέπει να είναι συνολικός αυτός ο διαχωρισμός, να απαγορεύεται να αναλαμβάνει τις δύο διαστηριότητες ο ίδιος οργανισμός, να υπάρχουν μήπως απλώς ορισμένοι περιορισμοί και όπως είπα και πριν υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις από τα διάφορα κράτη ως προς την εφαρμογή του κανόνα αυτή του διαχωρισμού. Ο σημαντικότερος στόχος βέβαια θα ήταν να μην λάβουμε υπόψη μας μόνο τα διαρθωτικά στοιχεία του διαχωρισμού αυτού, αλλά η ιδέα ότι αυτό το ring fencing είναι κάτι το ουσιαστικό για την οικονομία και ότι οι δραστηριότητες αυτές και οι δύο δεν θα συμβάλλουν στην αύξηση της αστάθειας ή πιθανής αστάθειας και σε περίπτωση πτώχευσης της τράπεζας θα πρέπει να υπάρχει μια λύση που να μην βασίζεται μόνο στην δαπάνηση χρημάτων των φορολογουμένων. Είναι λοιπόν το θέμα αλλαγής νοοτροπίας, τραπεζικής νοοτροπίας. Ορισμένοι είπαν ότι η βασική δοκιμή, η ουσιαώδης δοκιμή για το διαχωρισμό ή ring fencing θα ήταν η αλλαγή νοοτροπίας. Δηλαδή η νοοτροπία που δέχεται την ανάληψη υψηλού κινδύνου από τις τράπεζες έχει καταλήξει σε αρνητικά αποτελέσματα και επομένω πρέπει να δούμε ποιες είναι οι βασικές τραπεζικές δραστηριότητες που είναι η αποδοχή καταθέσεων και η δανειοδότηση χωρίς ανάληψη υψηλού κινδύνου. Πρόσθε, επιπρόσθετα, στις προτάσεις Λίκανεν πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις. Γιατί βρέπουμε τα πράγματα πολύ βραχυπρόθεσμα με μόνο γνώμονα το κέρδος. Πρέπει λοιπόν να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά και να βασιστούμε περισσότερο το θέμα του συνδυασμού όλων των τραπεζικών δραστηριοτήτων με το σύνολο της πραγματικής οικονομίας. Η δανειοδότηση των ε, κολαπτωμένων επιχειρήσεων είναι κάτι πολύ ουσιαστικό και πρέπει να ζητήσουμε, να αποζητήσουμε προτάσεις για να μπορέσει να υπάρξει δανειοδότηση για ανάπτυξη. Υπάρχουν και θέματα ανταγωνιστικότητας βέβαια. Τα τελευταία δέκα χρόνια δεν ιδρύθηκε καμία καινούρια σημαντική τράπεζα. Οι πελάτες συνεχίζουν να ζητούν περισσότερο δίκαια μεταχείριση και καλύτερη απόδοση βέβαια και υπάρχουν ήδη ενδείξεις αλλαγών, μιας επανάστασης στην τραπεζική διαχείριση. Υπάρχουν νέες ιδέες όπως το peer-to-peer -peer lending Ξέρουμε ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση. 14 τεράστιες τράπεζες τα ελέγχουν όλα, 15 τράπεζες ελέγχουν 54% της αγοράς και αντιπροσωπεύουν 150% του ενωσιακού ΑΕΠ. Ο λόγος τραπεζικού μεγέθους με το ΑΕΠ έχει τριπλασιαστεί Άρα η ανταγωνιστικότητα είναι απαραίτητη για να υπάρχει σωστός τραπεζικός τομέας. Πρέπει να υπάρξει όμως μεγαλύτερη διαφοροποίηση και τραπεζική λειτουργία που να στοχεύει περισσότερο τον καταναλωτή και αυτό φυσικά θα βοηθήσει εκ νέου και αυτό την πραγματική οικονομία. έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν πιο εύκολα να αλλάξουν τράπεζα ή δραστηριότητα. Τελειώνω με κάτι καινούριο που συνέβη, σημειώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Handelsbanken ανοίγει κάθε δύο εβδομάδες νέο υποκατάστημα διαχειρίζεται υποθήκες και χορηγεί μικρά, μικρού επιχειρησιακά δάνεια, δεν πληρώνονται πριν στους υπαλλήλους της και γενικά λειτουργεί πολύ καλά. Οι καταθέσεις επενδύονται από τους ιδίους τους υπαλλήλους της τράπεζας και των πελατών και επομένως πρέπει να υποστηρίξουμε τέτοιου είδους τράπεζες που ακολουθούν διαφορετικό τραπεζικό πρότυπο, διαφορετική νοοτροπία που είναι κάτι νομίζω τελείως απαραίτητο μακροπρόθεσμα, όχι βραχυπρόθεσμα μόνο για μπαλώματα αλλά να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη λύση και αλλαγή. Και έχουμε εδώ την ευκαιρία με την έκθεση Λίκανεν να επιμείνουμε σε αυτό. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις και των σκιωδών και υπολείπων συναδέλφων και θα καταθέσω στην επόμενη εβδομάδα την πρότασή μου Απλώς σήμερα ήθελα να ακούσετε μερικές καινούργιες ιδέες και επαναλαμβάνω θέλω να ακούσω τις απόψεις σας. Ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αρλίν, για τις ενδιαφέρουσες ιδέες. Θα ακούσουμε πρώτα τους Σκιώδης Κάρεν, για το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αρλίν για την ε, η περιστατωμένη επεξεργασία των βασικών στοιχείων της έκθεσης Λικάνεν, καθώς και κάποιων πρόσθετων ιδεών που έθεσε επιτάπητος, που σίγουρα θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση και πρέπει να συμμετέχουμε γιατί η συζήτηση για την έκθεση Λίκανεν και για την διαπτωτικές αλλαγές του τραπεζικού τομέα συμπληρώνουν τις μεγάλες τις σπουδές νομοθεσίες που πέρασε το Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια και που είναι τώρα σε εφαρμογή. Γι' αυτό και η πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω αφορά ότι αυτό το μεγάλο πακέτο, το νομοθετικό πακέτο που αυτή τη στιγμή συζητείται και τίθεται σε εφαρμογή, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ε, το ποιο, ποια στάση θα κρατήσουμε. Ε, η στάση αυτή να είναι αρκετά στεναρή όσον αφορά την προστιθέμενη αξία σε σχέση με αυτή την νομοθεσία και τις συνεχιζόμενες αλλαγές που προκαλούνται από αυτήν. Θα πρέπει να είμαστε επίσης αρκετά στεναροί ώστε να σχετιζόμαστε με τη ε, το γενικότερο μας στόχο, δηλαδή την ε, μεγαλύτερη ασφάλεια στις τράπεζες. Γι' αυτό και αυτή εδώ είναι μια δοκιμασία για να δούμε τι θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε οικονομική σταθερότητα και πιο υπεύθυνη ε, συμπεριφορά όσον αφορά την ανάληψη κινδύνων. Θέλουμε επιστροφή της εμπιστοσύνης στη διατραπεζική αγορά και την αποκατάσταση των γραμμών των πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία. Θέλουμε διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τις τράπεζες και αυτό είναι κρίσιμο θέμα και θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη βεβαιότητα των τραπεζικών μοντέλων. Έχουμε μικρές και μεγάλες τράπεζες στην Ευρώπη και αυτό διαφοροποιεί την βάση. Το να διατηρήσουμε διεθνή πρότυπα επίσης ναι, είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό πιστεύω πως είναι επίγονο να διατυπώσουμε μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή σε σχέση με τις διαθετικές μεταρρυθμίσεις. Γιατί όπως είπε σωστά Αρλίνα, έχουμε την έκθεση Λίκανεν, Έχουμε διάφορους άλλους κανόνες, αλλά όταν συγκρίνουμε την προσέγγιση Λίκανεν με την ε, προσέγγιση Φίκερ, σε αυτήν το λιανικό κομμάτι των τραπεζών είναι ξεχωριστό και υπόκειται σε περισσότερες κεφαλιακές απαιτήσεις, ενώ στην προσέγγιση Λίκανεν το εμπορικό τμήμα χωρίζεται και υπόκειται σε μεγαλύτερες κεφαλαϊκές απαιτήσεις. Τι σημαίνει αυτό, αν ε, αρχίσουμε και κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση όπου οι περισσότερες τράπεζες έχουν παραδείγματα στο Λονδίνο αλλά και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αν ακολουθήσουν αντίθετη προσέγγιση και είναι δυνατόν και αυτό θα το προτιμούσαν να έχουμε ένα είδος ε, σύνθεσης μιας κοινή προσέγγισης που να είναι ο στόχος μας. Πιστεύω πως σωστά ανέφερες ε, πάρα πολλά ζητήματα σε σχέση με την επιλογή που προτείνει η έκθεση Λίκανεν για το πώς ναι. ορίζεται το εμπόριο ιδιοκτησίας ποιος, ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής, αν θέλουμε να περιχαρακώσουμε, να έχουμε νομική διαχωρισμό, ε, αυστηρό διαχωρισμό και θέτω όλα αυτά τα ερωτήματα επιτάπητος γιατί πρέπει να τα εξετάσουμε. Δεν έχω απόλυτα ξεκαθαρίσει τι πρέπει να κάνουμε εδώ, αλλά και είμαι ανοιχτή συζήτηση και βεβαίως θα δούμε και ποια θα είναι η διάθεση όλων προς, αυτή την κατέ, προς τις δικές μου ε, ε, προτάσεις. Να πω και δύο λόγια για την διακυβέρνηση σε σχέση με το θέμα της ε, διάλυσης ή της εξαγοράς θα το συζητήσουμε αργότερα αλλά θα πρέπει για να, να αλλάξει η νοοτροπία όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Αυτό που λείπει ωστόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ένας διάλογος στον ίδιο το τομέα, στον ίδιο το κλάδο ε, και ο νομοθέτη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα βελτιωθεί η διακυβέρνηση, πώς θα έχουμε πιο βιώσιμο τραπεζικό τομέα και εδώ και εκεί ίσως και να υπάρχουν τράπεζες που ε, προτείνουν κάποια πράγματα στην ε, κάτω χώρες έχουμε έναν κώδικα διοντολογία. επί τη βάση πολλών τέτοιων συζητήσεων φτιάχτηκε. Θα έπρεπε να έχουμε λοιπόν έναν ευρωπαϊκό κώδικα διοντολογία για τις τράπεζες και οι τράπεζες θα πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουν ότι όταν δεν υπάρχει επαρκής πρόοδο, η πιθανότητα να νομοθετήσουμε σε τομεί όπου θα προτιμούσε ο ίδιο ο κλάδο να έχει προτείνει βιώσιμε λύσει, θα έπρεπε να το κάνει. Νομίζω λοιπόν πως πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι εδώ και όχι ε, να κρατάμε αμυντική στάση. Δείτε τι έγινε με το πεδίο των κεφαλαικών απαιτήσεων και των αμοιβών. Ε, εμείς θα πρέπει να εμπιστευτούμε και τον ίδιο τον κλάδο για να κάνει πιο βιώσιμες προτάσεις και να αλλάξει και την νοοτροπία του. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου για την ώρα και προσβλέπω σε περαιτέρω συζήτηση εδώ στην Επιτροπή και με τους κοιόδες εισηγητές και με εσά ως εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Äh, Ευχαριστώ Σάρων και Αλέν για την έκθεση. Φαίνεται πως έχετε κάνει ένα καλό κείμενο και αναμένουμε και τη γραπτή έκδοση. Για τους στόχους συμφωνούμε όλοι. Θέλουμε περισσότερη σταθερότητα στο τραπεζικό τομέα, ελάφρυνση του φορολογούμενου, οι τράπεζες να ασχοληθούν με την κύρια δουλειά τους, δηλαδή χρηματοδότηση της πραγματικής ε, οικονομίας και αλλαγή νοοτροπίας. Αλλιώς δεν θα έχουμε αλλαγή. Ενδιαφέρον είναι πως παρά το ότι συμφωνούμε από την Αμερική έως την Ευρώπη, ε, ενδιαφέρουν ε, κατά πολύ οι αναλύσεις μας. Στην Αμερική πιστεύουν, Mr. Φόλκ και οι λοιποί, πως έφταιγαν οι, traders ε, για αυτό το θέμα και πρέπει να περιοριστούν. Βεβαίως ε, το πόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτό δείχνει, ε, πόσο, το δείχνει το πόσο αργά εφαρμόζονται οι προτάσεις τους γιατί και ο ορισμός του τι είναι spot trading και market making δεν είναι τόσο εύκολη. Γι' αυτό έχουμε εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται μια πρόταση η οποία δεν θα περάσει. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε κάτι το απλούστερο, το τι είναι λιανική και το να, πώς μπορεί να απομονωθεί Οπότε αυτό το οποίο με λυπεί είναι πως ε, κάποιες χώρες, ε, η Γαλλία, η Γερμανία, ε, Ηνωμένο Βασίλειο, αντί να συνεννοηθούν να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα, σπέβδουν να κάνουν δηλώσεις ότι δεν θα έχουμε μια ευρωπαϊκή λύση, αλλά πολλές εθνικές τροποποιήσεις, κάτι το οποίο βεβαίως δεν μας βοηθά. Γιατί μετά έχουμε το πρόβλημα πως δεν θα έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού στην αγορά. Η πρόταση Λικάνεν να μην ε, δούμε μόνο την, ε, τις κινήσεις που κάνει η διατραψά και, το market making συνολικά νομίζω πως θα πρέπει να δούμε το τι θα γίνει στην πράξη για να το κρίνουμε ο κλάδος και μάλιστα όχι μόνο οι εκπρόσωποι των τραπεζών που κάνουν όλες τις εργασίες αλλά και των λοιπών τραπεζών ε, είναι κάπως επιφυλακτικοί. Ε, επίσης είναι θετικό το ότι γίνονται προτάσεις για την διάσωση και τυχόν κλείσιμο ε, των τραπεζών και βλέπουμε παραδείγματος χάρη στο παράδειγμα της Ολλανδικής Τράπεζας SNS. Πώς βραχυπρόθεσμα δεν γλιτώνουμε τη συμμετοχή του φορολογούμενου όταν ε, έχει μεγάλες δυσκολίες μια τράπεζα. Δυστυχώς ε, παρόλες τις προτάσεις ε, και σε όλες τις προτάσεις που υπάρχουν η πραγματικότητα είναι πως θα πρέπει να πληρώσει ο φορολογούμενος αν και στην περίπτωση της SNS ε, πλήρωσαν και οι ε, μετοχοί. Είχαμε ένα bail-in δηλαδή. Αυτό το οποίο με ενοχλεί είναι ε, πως έχουμε μία πρόταση Λικάνεν και βεβαίω βασιζόμαστε σε μια έκθεση ιδέα πρωτοβουλία και η Κομισιόν, από ό,τι φαίνεται, πριν το καλοκαίρι θα καταθέσει μια νομοθετική πρόταση, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την διαχείριση της κρίση τρέχουσα. Οπότε εργαζόμαστε σε διάφορα μέτωπα και θα πρέπει βεβαίω να δούμε και τα αποτελέσματα των διαφόρων αυτών ε, δράσεων. Και ελπίζω να καταλήξουμε σε κάτι ομοιόμορφο. Αυτό το οποίο ε, πρέπει να συζητήσουμε για το μέσο Μπέιλιν ε, είναι το ποιος θα πρέπει να, να συμπεριλαμβάνεται σε αυτός. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν μπορεί να αγοράζει το μέσο Μπέιλιν ε, συμμετοχής ε, των ε, μετόχων μια άλλη τράπεζα. Γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να συμπεριληφθεί μια τέτοια επισφάλεια στους λογαριασμούς μιας τράπεζας. Αλλά εάν είναι βεβαίως αν έχουμε τη συμμετοχή συνταξιδοτικών ταμείων κτλ. πάλι ποιος πληρώνει ο φορολογούμενος ή ο συνταξιούχος μέσω κάποιου τρίτου βεβαίως. Δεν ξέρω λοιπόν ποιος θα έπρεπε να είναι ο ιδεώδης επενδυτής για αυτό το μέσο Μπέιλιν. Για το θέμα τώρα της ε, διακυβέρνησης, συμφωνώ με αυτό το οποίο είπες εσύ και οι προλαλήσαντες και η Κάριν. Είναι λυπηρό το ότι ο κλάδος δεν προσπαθεί με βάση τα όσα πήγανε ήδη στραβά από μόνος του να κάνει κάποιες λογικές προτάσεις και να μας δώσει το μήνυμα πως ναι εντάξει παραδεχόμαστε πως πήγαν κάποια πράγματα στραβά, θέλουμε να τα κάνουμε καλύτερα στο μέλλον. Ανταυτού εξακολουθούν να αμήνονται και να διατηρήσουν, να θέλουν να διατηρήσουν το status quo. Ανθρώπινο και κατανοητό, γιατί κανείς δεν θέλει αλλαγή, αλλά είναι και πραγματικά ε, εσχρό από την άλλη. Ευχαριστώ πράσινη τώρα, Φιλίπ. Ευχαριστώ Σάρον. Νομίζω πως ε, έχουμε τους ίδιους στόχους. Θα ήθελα να τονίσω δύο από αυτούς. Ο ένας είναι να μειωθεί η υπερβολική δύναμη κάποιων τραπεζών, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Μου προξενεί εντύπωση το ότι ένα μικρός αριθμό μεγάλων τραπεζών έχουν κυριαρχία στην τράπεζα λόγω αυτής της ε, ε, υπονοούμενης, αν θέλετε, εγγύησης. Οπότε θα πρέπει να αποκατασταθεί ο ανταγωνισμός. Δεν είναι φυσιολογικό κάποια ιδρύματα να μπορούν να χρηματοδοτούν δραστηριότητε με καλύτερους όρους, πιο ευνοϊκούς όρους, γιατί έχουν την υπονοούμενη αυτή, αν θέλετε, εγγύηση των, των φορολογουμένων. Να πω κάποια πράγματα τα οποία ακούγονται από τον κλάδο και από, τους, ε, από τα φερέφωνα των τραπεζών. Κοιτάξτε, να σας πω εγώ που ζω στο Βέλγιο και μιλάτε για στις τράπεζες. Οι τράπεζες ήταν γενικές τράπεζες, έκαναν όλες τις εργασίες και ακριβώς χρεοκόπησαν γιατί δεν υπήρχε διαχωρισμός μεταξύ των όσων έκαναν στις χρηματαγορές, κυρίως subprime, και του τι έκαναν ως λιανικές τράπεζες. Γι' αυτό έπρεπε να τις διασώσουμε. Εάν υπήρχε διαχωρισμός, δεν θα χρειαζόταν να πάμε στην διάσωση της Φόρτης, Δέξια, Καμπεσέ και λοιπόν. Και το Βέλγιο δεν είναι μοναδική περίπτωση, οπότε δεν είναι αλήθεια πως είναι πιο εύρωστο το μοντέλο των γενικών τραπεζών. Έχουν χρεοκοπήσει γενικές τράπεζες, επενδυτικές τράπεζες, τράπεζες λιανικής, οπότε πρέπει να υπάρχουν όρια μεταξύ των δραστηριοτήτων. Μετά, οικονομίες κλίμακας. Αυτό ισχύει ε, ως ένα βαθμό. Μετά, όσο αυξάνεται ε, το μέγεθος, συμβαίνει το αντίθετο. Ε, είναι πιο ακριβό, εάν όχι αδύνατον, να διαχειριστούμε τράπεζες του μεγέθου της Deutsche Bank, Barclays και λοιπόν. Επίσης, ε, όλοι, λέτε πως όλοι οι πελάτες θέλουν ε, να ασχολούνται και να συναλλάσσονται με μία τράπεζα. Εγώ εργαζόμουν σε πολύ μεγάλη εταιρεία πληροφορικής που έκανε τα πάντα. Κανείς πελάτης μας δεν ήθελε να αγοράσει τα πάντα από μας. Γιατί? Γιατί ήθελε να δημιουργήσει ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών. Δεν, δεν στέκει λοιπόν αυτό. Μετά λέτε Πώ εάν είμαστε πάρα πολύ σκληροί θα πάνε στη σκιώδη τραπεζική. Ίσως υπάρχει κάποιο τέτοιο ρίσκο. Αλλά γι' αυτό η Κομισιόν θα καταθέσει προτάσεις να το αντιμετωπίσει. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ελέγχου στα όρια, αν θέλετε, στα σύνορα μεταξύ σκιωδών τραπεζών και τραπεζών. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να τζογάρει κανείς τα δικά του λεφτά και να τα χάνει ή να απολαμβάνει τα κέρδη. Κανένα πρόβλημα. Αρκεί όχι ε, κορώνα κερδίζω γράμματα χάνεις όμως. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Και μετά μας λέτε πως θα καταστραφούν θέσεις εργασίας. Ε, ένα από τα δύο θα γίνεται. Ή θα λέτε πως υπάρχουν οικονομίες κλίμακας. Δηλαδή οικονομίες κλίμακας σημαίνει πως καταργείς δουλειέ. Και μετά μας λέτε άμα διαχωριστούν οι τράπεζες θα μας λέτε πως θα χάθουν πάλι δουλειές. Ε, ε, τι, ή το ένα ή το άλλο. Δεν μπορεί να τα, να τα λέτε και τα δύο μαζί. Αυτό που θεωρούμε είναι πως εάν γίνουν μικρότερα τα τραπεζικά ιδρύματα θα δημιουργηθούν δουλειές αντί για το αντίθετο. Μετά, η δημιουργία αγορών είναι ουσιαστική για την ε, οικονομία. Εμεί δεν είπαμε να μην υπάρξει τέτοια δημιουργία αγορών, αλλά οι δραστηριότητες αυτές να τιμολογούνται σε τιμές αγοράς. Να μην ευνοούνται σε κάποια ιδρύματα από την ε, επιδότηση αυτή η οποία υπονοείται. Και είχαμε μια συζήτηση της ε, προάλλης και μας ρώτησε ο ΜΑ. ρωτήσα μάλλον ε, ξεκάθαρα τον εκπρόσωπο της Deutsche Bank από ένα Υπουργείο Οικονομικών και τον ρώτησαν, πείτε μας, ναι ή όχι, συμφωνείτε πως το τραπεζικό σας ίδρυμα πρέπει να πληρώσει τιμή αγοράς για τις δραστηριότητες του στις χρηματαγορές, δηλαδή τιμή η οποία δεν θα λαμβάνει υπόψη την υπονοούμενη αυτή επιδότηση της διάσωσης από το φορολογούμενο. Και μας απάντησε όχι. Μας είπε η Deutsche Bank δεν θέλω να πληρώσω την πραγματική τιμή ε, των δραστηριοτήτων μου στην αγορά. Α, εντάξει, αυτά. Μέχρι εκεί φτάνει η οικονομία της αγοράς. Δηλαδή καμιά φορά αισθάνομαι πως είμαι ο μόνος φιλελεύθερος εδώ μέσα. Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι η αγορά των ε, παραγωγών έχει μέγεθος 11 φορές την πραγματική οικονομία. Κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει και κάποια ε, κάποιος συσχετισμός και κάλυψη αυτής της αγοράς. Δεν νομίζω να χρειάζεται τόσο μεγάλο μέγεθος. Τέλος, για την ευρωπαϊκή σε σχέση με την εθνική προσέγγιση. Λυπούμε για το ότι έχουμε εθνικές προσεγγίσεις, αλλά θα πω το εξής. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε και ζήτησε μία ανεξάρτητη ε, επιτροπή για τις ε, τράπεζες, δεν θα γινόταν τίποτα και χρειάστηκε καιρό η Κομισιόν να αναγνωρίσει πώς χρειάζεται κάτι. Αλλά η διαδικασία έχει ξεκινήσει από πριν. Αυτό το οποίο εγώ δεν καταλαβαίνω είναι πως και το Βερολίνο και το Παρίσι τώρα πάνε προς κάποιες χλιαρές μεταρρυθμίσεις ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πως κάτι γίνεται ήδη. Γι' αυτό θεωρώ αυτές τις πρωτοβουλίες μια προσπάθεια να προκαταλάβουν σοβαρές μεταρρυθμίσεις της Επιτροπής μας. Γι' αυτό στην τέταρτη οδηγία κεφαλαιακών απαιτήσεων είχαμε ομόφωνη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την ΚΟΕ μέχρι τους συντηρητικούς και παραπέρα για κάτι τόσο κρίσιμο όπως τράπεζες. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να το επαναλάβουμε αυτό το κατόρθωμα και στο προκείμενο εδώ πέρα θέμα. Γιατί θεωρώ πως υπάρχει πολύ μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων που θέλουν πραγματικά οι τράπεζες να εξυπηρετούν την πραγματική οικονομία. Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε και έτσι θα ισχυροποιηθούμε και μελλοντικά στι διαπραγματεύσει. Αλλά θα είναι βλαβερέ διαπραγματεύσει όχι μεταξύ ημών, αλλά μεταξύ ημών και των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Οπότε περνάμε τώρα στο ECR και πέρα από το ECR. Ο κ. Καμολέβα, θέλετε να σας τα πω και αυτά και τα άλλα, αν θέλετε να αναλάβω αυτό τον όρο τον ρόλο με συγχωρείτε. Καταρχήν, όπως και άλλοι σε αυτή την επιτροπή, να σας πω ότι μετά πέντε χρόνια από την πρώτη κρούση στο Ηνωμένο Βασίλειο πάνω από τέσσερα χρόνια μετά από την Lehman Brothers έχουμε μια ε, νομοθεσία ε, στεναρή αλλά δεν έχουμε αντιμετωπίσει το βασικό πρόβλημα ότι δηλαδή αν αύριο μια τράπεζα ε, πτώχευε πάλι θα ήθελε οι φορολογούμενοι να πληρώσουν τα σπασμένα. Ε, αυτό είναι το βασικό και πρέπει να πούμε όσο γίνεται, ακόμα και αν είναι δύσκολο, ότι όταν μια, τρα... μια κυβέρνηση έχει την εξουσία, δεν ε, θα πρέπει πια οι φορολογούμενοι να πληρώσουν τα σπασμένα και υπάρχει στήριξη γι' αυτό. Θέλουμε οι αγορές να δουλεύουν. Γιατί τα αποτυχημένα θεσμικά όργανα να πληρώνονται από τους φορολογούμενους. Ενώ οι αριστεροί λένε γιατί τους θα δώσετε ε, τα χρήματα των φορολογούμενων σε αυτές τις πλούσιες τράπεζες. Υπάρχει όμως συνένεση τελικά παρότι είμαστε από αντίθετα πολιτικά φάσματα να διαφωνούμε με την χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για το κλείσιμο τραπεζών. Δηλαδή να, να, να, Συνεχίζουν όμως να λειτουργούν τα ATM, να συνεχίζει ο κόσμος να μπορεί να πάρει τα χρήματά του, γιατί διαφορετικά θα υπάρξει κοινωνική ε, αταξία και ε, πρόβλημα. Πρέπει να ξεφύγουμε λοιπόν από αυτή την ιδέα του ότι είναι πολύ μεγάλα για να καταρρεύσουν ε, κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όταν μιλά κανεί με διάφορε τράπεζε, ε, παίρνει διαφορετικέ απαντήσει. Ε, κάποιο διευθύνων, κάποιο υψηλά ιστάμενο μια Βρετανική Τράπεζα, μου είπε ότι δεν είμαστε ακόμα αρκετά καλοί στο να συνομιλούμε μεταξύ μα. Ενώ ένα εκπρόσωπο μια Αυστρικής Τράπεζα, μου είπε «Συγγνώμη, μα είναι πολύ μεγάλε κάποιε τράπεζε για να καταρρεύσουν». Μα και εγώ είπα συγγνώμη, μα δεν γίνεται έτσι. Και ενώ εκπρόσωπο κάποιες γερμανική τράπεζα μου είπε, Μα εσεί νομίζετε πω μα αρέσει να μα εγκλητώνουν τα χρήματα των φορολογούμενων. Ναι, εντάξει όλα αυτά. Αλλά μετά τι κάνουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε στην πράξη. Πρέπει να βρεθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Έπειτα, άμεση ευθύνη. Εάν κάτι το οποίο επίσης μας ενώνει σε όλο το πολιτικό φάσμα είναι ότι κανείς δεν ανέλαβε πραγματικά ευθύνη για την κακή διαχείριση της τράπεζάς του. Και θα ήθελα λοιπόν να εστιάσουμε την προσοχή στην άμεση ευθύνη. Ποιο είναι άμεσα υπεύθυνο, πόσο μπορούμε αυτό να το, να το οθήσουμε ή να βρούμε κάποιο μέση εδώ ώστε να εξασφαλίσουμε πως οι διευθυντέ θα εκτίθεται ε, κάποιο άλλη πρόταση, εν περιπτώσει, ώστε κάποιο να πληρώσει το τίμημα. Δεν έχω πρόβλημα αν μια τράπεζα πάει καλά, εξυπηρετεί τους πελάτες της και κερδίζει, ο διευθυντή τη να κερδίζει πολλά χρήματα. Αλλά όταν αποτυχάνει, ε όχι πάλι να παίρνει μπόνους. Το ε, επόμενο θέμα είναι τα πρότυπα τα λογιστικά. CDO, CDS, θα βάλουμε και αυτά, ιδιαίτερα οι επενδυτικές τράπεζες, όχι οι τράπεζες ε, οι άλλες. Το θέμα είναι όμως αν αυτό σκάσει, τότε η τράπεζα να έχει τα χρήματα στην άκρη. Να έχει αυτό που λέγαμε lost provision και prudence. Να έχει τα χρήματα στην άκρη για να πληρώσει την έκθεσή της και την απώλειά της, τη ζημιά της. Τρει δολάρια είχε εκτεθεί η AIG. Ε Μα πώς θα μπορούσε ποτέ να πληρώσει γι' αυτά. Και τα λογιστικά πρότυπα του επέτρεπαν να το κάνουν αυτό, γιατί φύγαμε μακριά από την πρόληψη και από την πρόνοια. Θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα να βάζει κανεί τα χρήματα στην άκρη για δυνητικέ απώλειε. Έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα που δεν δηλώνει κανεί την απώλειά του παρά μόνο όταν πια την έχει δει. Έχουμε επιτρέψει τα λογιστικά στάνταρ να προχωρήσουν κατά προς αυτή την κατεύθυνση και πολλοί κόσμοι μου είπαν, όπως δεν εμπιστεύεται τα ισοζύγια των τραπεζών, τους ισολογισμούς και ότι θα πρέπει να προχωρούν σε ανάλυση ε, βαθύτερη των τραπεζών. Και κάτι ακόμα όσον αφορά τον έλεγχο. Και πάλι πολύ μεγάλος προβληματισμό όσον αφορά ε, τον έλεγχο που έχει φτάσει σε μια κατάσταση όπου οι ελεγκτές δεν ελέγχουν, δεν αμφισβητούν την Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας και να τους πει γιατί εκεί είναι πιο ψηλός ο αριθμός και εκεί πιο χαμηλός. Λένε απλά μην ανησυχείς, έχεις κάνει σωστά τη διαδικασία, βάζουμε το OK και προχωράμε. Και μετά βλέπουμε ένα σωρό τράπεζες να καταραίουν μετά, ε, ενώ έχουν πάρει το σιχωροχάρδι από τον έλεγχο, τον λογιστικό. Επίσης, ο περισσότερος κόσμος πιστεύει πως τα χρήματα το καταθέτει και μένουν εκεί, στην τράπεζα. Στην ουσία όμως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι δανείζουν τα χρήματά τους στην τράπεζα και εκείνη τα χρησιμοποιεί. Θα έπρεπε ωστόσο ο καταθέτης να γνωρίζει τι κάνει με την, η τράπεζα με τα χρήματά του. Και ίσως να υπάρχει και ευκαιρία να υπάρχει ένας ε, λογαριασμός κατάθεσης ε, Μπορεί να μην έχεις, ε, να μην έχεις ε, επιτόκιο, αλλά τουλάχιστον ξέρεις πως τα χρήματα αυτά είναι εκεί, τα προσέχει κάποιος και ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το θα θες εσύ θα τα, θα τα πάρεις πίσω και να μην εξαρτάσει μόνο από τα προγράμματα εγγύησης, καταθέσεων κτλ. Απλές ιδέες, ας πούμε. αλλά αν τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα εξ αρχής, ίσως να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Νομίζω πως ε, έχουμε κοινέ απόψεις με την ησυχήτρια και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί της και με τους υπόλοιπους σκιώδης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελείωσε ο γύρος των σκιωδών. Θα μιλήσουν τώρα οι απλοί συνάδελφοι. υπερβάνς προς το τέλος και η Κομισιόν είναι εδώ παρούσα. Δεν ξέρω αν έχει κάτι να μας πει. Άλλα σύντομα όλοι, γιατί έχουμε μόνο 10 λεπτά θεωρητικά. Ολύν, Λίαμ. Ευχαριστώ Σάρον. Ευχαριστώ και την Αρλέν γιατί περιέγραψε σωστά τα δεδομένα του προβλήματος. Η έκθεση Λικάν είναι πολύ σημαντική γιατί η τραπεζική μεταρρύθμιση ίσως είναι η μεταρρύθμιση που θα ολοκληρώσει την τραπεζική ένωση που λένε. Είναι κάτι που και οι Αμερικανοί δεν το έχουν ακόμη τολμήσει. Και γι' αυτό είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν να καθορίσουν τους κανόνες του παιχνιδιού, γιατί σήμερα υπάρχουν χώρες που προδικάζουν τα αποτελέσματα, προτρέχουν και έχουν εφαρμόσει τμηματικές μεταρρυθμίσεις, είτε γιατί πιέζονταν από ορισμένα λόμπι, είτε γιατί τα, είχαν τα εθνικά τους συμφέροντα που τους ανάγκαζαν να μην προχωρήσουν περαιτέρω. Πρέπει να καθοριστεί λοιπόν το γενικότερο πλαίσιο. Δύο θέματα μου φαίνονται σημαντικά εδώ. Πρώτον, η περίμετρος των κερδοσκοπικών λεγόμενων δραστηριοτήτων που πρέπει να πλαισιωθούν και υπάρχουν πολλοί ορισμοί για αυτές. Η καλύτερη είναι της έκθεσης Λίκανεν που περιλαμβάνει 16% των δραστηριοτήτων των τραπεζών. Υπάρχει και γαλλική νομοθεσία που μιλάει μόνο για 1% των κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων που θα πλαισιώνονται. Μεταξύ του 1% της Γαλλίας και του 16% του Λίκανεν νομίζω μπορεί να βρεθεί το σωστό όριο. Ξέρουμε ας πούμε ότι μόνο 7% των κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό ιδιαίτερα. Δεύτερο θέμα, η φύση του διαχωρισμού. Στην έκθεση Λίκανεν προτείνεται να ληφθούν υπόψη οι θυγατρικές, οι δραστηριότητες των θυγατρικών, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύουν στις επενδυτικές τράπεζες άλλη δραστηριότητα. Πρέπει λοιπόν και εμείς να δούμε πώς θα γίνει ο διαχωρισμός. Θέλουμε να διατηρήσουμε τον ομφάλιο λόρο μεταξύ των κύριων δραστηριοτήτων και ή των δραστηριοτήτων της κύριας τράπεζας και της ιατρικής της που θα ασχολείται με τις επενδύσεις ή όχι. Ή θα κάνουμε πλήρη διαχωρισμό. Εδώ τίθενται τρία προβλήματα. Ένα, η ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες. Αν δεν υπάρξει σαφής διαχωρισμός, τότε θα παραμείνει αυτή η γελία έννοια του too big to fail. Και θα πληρώνουν πάντα οι φορολογούμενοι, εφόσον μιλάμε για κρατική εγγύηση. Και αν δεν κάνουμε το διαχωρισμό, τότε το πρόβλημα είναι ότι θα υπάρχει αυτή η έμεση κρατική εγγύηση και θα χρειάζεται να διασωθούν όλες οι δραστηριότητες της τράπεζας, όχι μόνο οι κύριες. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να την και να ενθαρρύνουν την Επιτροπή μας να προχωρήσει δυναμικά εδώ πέρα είναι η σημαντικότερη και ίσως η τελευταία μας ευκαιρία σε αυτή την θητεία να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα που έχει μεγάλη σημασία για τους ψηφοφόρους μας και να δείξουμε πραγματικά το τι πιστεύουμε. Πρέπει να δούμε το θέμα ευρύτερα όχι μόνο ως απάντηση στην έκθεση Λικάνεν, αλλά το είπαν ήδη κάποιοι συνάδελφοι, να ασχοληθούμε όχι μόνο με τις μεγάλες τράπεζες και το too big to fail, αλλά και τον διαχωρισμό με αυτό το οποίο λέμε σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Σε αυτό αναμένουν απαντήσεις οι ψηφοφόροι. Επίσης, να υπενθυμίσω πως εδώ και χρόνια λένε πως πρέπει να ελέγχεται κάθε φορέας, κάθε ε, οικονομική δραστηριότητα. Γιατί έχουμε το πρόβλημα του ότι κάνουμε πάρα πολλές τεχνικές εκθέσεις. Εντάξει δεν γίνεται διαφορετικά, αλλά ακριβώς αυτή η έκθεση νομίζω είναι μια μεγάλη ευκαιρία και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω σε αυτό να κάνουμε το εξής. Γιατί ε, πρέπει να πούμε πως δεν είναι σύμπτωση πως ε, αυτοί οι οποίοι υπερασπίζονται το City του Λονδίνου πάλι απουσιάζουν σήμερα και δρούν ως άμεση λομπίστες αυτών των μεγάλων τραπεζών και δεν είναι ε, δυνατόν μόνο να λένε πως εκπροσωπούν τους πολίτες αλλά είναι και ένας παράλογος εθνικισμός του UKIP και πρέπει να τα πούμε αυτά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω. Νομίζω πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν το κάνουμε αυτό να μην είναι το καλύτερο εχθρός του καλού. Αν δείτε τι έγινε με τον κανόνα Βόλκερ στις Ηνωμένε Πολιτείε. Μια απλή ιδέα δηλαδή που έγινε πάρα πολύ περιπλοκή με το να προσπαθήσουν να ορίσουν ακριβώς το τι θα έπρεπε να είναι στην κάθε γραμμή του κάθε ορίου. Και βεβαίω το όριο είναι κάπως θολό. Οπότε χοντρικά με το δούμε δεν έχει σημασία που θα πάει ένα 5% των δραστηριοτήτων. Σημασία έχει το 95% το οποίο πρέπει να διαχωριστεί. Οπότε πρέπει να δούμε την επάρκεια κεφαλαίου και τα σχέδια διάλυσης. Ε, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε σε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα είναι ακριβώς ενοποιημένο. Δηλαδή, εάν έχουμε ένα το αν θέλετε, σειρματόπλεγμα και ηλεκτροφόρο, σημασία έχει να μην υπάρχει, όπως είπα, να μην είναι διαπερατό. Τώρα το πού θα βρίσκεται ακριβώ είναι συζητήσιμο. Μπορούμε λοιπόν να το δούμε ευρύτερα. Όταν είχαμε την συζήτηση με τους Βόλκερ και Φίκερ ε, στο σεμινάριο του Φιλίπ και λοιπόν, εγώ κατέληξα να σκεφτώ πως ε, αυτό το οποίο προέκυψε είναι πως τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα εάν δεν τα κάνουμε απλά. Γιατί χωρίς απλοποίηση ναι. δεν ε, θα φτάσουμε στις λύσεις που τελικά θέλουμε. Οπότε νομίζω όλα εκεί περιέχονται. Το άλλο σχόλιο που θα έκανα αφορά τη συμμετοχή στις, διαδόσ, διασώσεις των μετόχων. Και οι επενδυτέ βεβαίως ε, δεν τρελαίνονται για κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει πως ε, θα πρέπει ίσως να υπάρχουν μεγαλύτερες αποδόσεις ε, γιατί τι θέλουν, θέλουν πάλι το κέρδος από ένα μέσο που αφορά τη χρεοκοπία μια τράπεζα χωρί να έχουν το ρίσκο. Δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή ιδέα, αλλά αν μία από τις συνέπειες ε, του μέσου αυτού είναι πως θα αρχίσει να κοιτάει την ανισότητα που υπάρχει μεταξύ της επένδυσης στο χρέος και της επένδυσης στο μετοχικό κεφάλαιο και βεβαίως σε κάποιους αρέσει περισσότερο το μετοχικό κεφάλαιο και για τους ε, και δούμε και τα φορολογικά ωφέλη του μέσου του χρέους, τότε κάποιοι θα σκεφτούν θα επενδύσω ανταυτού σε μετοχικό κεφάλαιο και θα είναι θετικό αυτό. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες σκέψεις που έχω. Τώρα, η τελευταία μιλήτρια είναι η Περβάνος. Ευχαριστώ, Σάρων. Θέλω να κάνω πολλέ παρατηρήσει. Καταρχήν, θέλω να ενθαρρύνω την Αρλίν, γιατί νομίζω πω η έκθεσή τη θα είναι πολύ ε, σημαντική. Πρώτο θέμα είναι το χρονοδιάγραμμα και ο χρόνο. Το θέμα της, ε, του διαχωρισμού των τραπεζικών δραστηριοτήτων, ειλικρινά, ορισμένοι άρχισαν να το συζητούν από τον Φθινόπορο του 2007. Ήταν τμήμα των επιτάπητων προτάσεων. Ε, και έκτοτε είμαστε τώρα σε μια φάση όπου φοβούμε πως αυτή η θητεία θα τελειώσει χωρίς το Κοινοβούλιο να έχει λάβει απόφαση πέρα από την έκθεση της Αρλίν για την πραγματικότητα και τελικά των όσων θα θεσπίσουμε για να τροποποιήσουμε την ε, τραπεζική δομή. Άρα λοιπόν τελικά είναι αρκετά κλασικό το παιχνίδι αλλά μπορεί εδώ να υπάρξουν ε, παράπλευρες ε, ε, επιπτώσεις που θα είναι αντίθετες. Τα πράγματα προχωρούν. Δεν ξέρω εσείς τι, τι, τι έχετε αποκομίσει από τα όσα γίνονται στην Γαλλία και ιδιαίτερα στην ομιλία του Μπουρζέ θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το θέμα ήταν ένα σημαντικό θέμα, κεντρικό θέμα της εκστρατείας στη Γαλλία. Υπάρχει μια δυσκολία και το βλέπουμε με βάση τα όσα ε, υιοθετούνται μέσα στο πλαίσιο της CRD4 τις οδηγίες για τις κεφαλαϊκές ε, απαιτήσει ε, και αυτό θα μας αναγκάσει να ξαναδούμε και την ομοθεσία που ναι. έχουμε σήμερα πια θεσπίσει. Ε, άλλη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι πέρα από τη διάκριση των δραστηριοτήτων ε, κατάθεσης και επενδύσεων της τράπεζας, των τραπεζών μάλλον, θα πρέπει να προσέξουμε να μην περάσει σιωπηρά το θέμα της δομής του τομέα του τραπεζικού το θέμα της αναλογικότητας, δηλαδή ανάμεσα στον τραπεζικό τομέα και την οικονομική δραστηριότητα μιας χώρας, όπως στην Ιρλανδία για παράδειγμα, για να αναφέρω μόνο αυτό το παράδειγμα, ή σε άλλα τραπεζικά πρότυπα, τα οποία επίσης μπορεί να ε, προκαλούν πρόβλημα είτε στο θέμα των καταθέσεων είτε στο θέμα των επενδύσεων. Τρίτη σειρά παρατηρήσεων. Ε, Πιστεύω ότι δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτές τις λύσεις όπου δίνουμε την εντύπωση ότι έχουμε απόλυτα ασφαλίσει τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας επειδή ξεχωρίσαμε τις καταθέσεις από τις επενδύσεις, διότι τότε θα αφήναμε τις επενδύσεις να αναπτυχθούν μέσα σε συνθήκες που δεν μπορούν να σταθούν από τη στιγμή που εξαρτάται από ένα μοντέλο το οποίο επίσης πρέπει να ε, πείσουμε με όσο γίνεται πιο μεγαλύτερη πεποίθηση, δηλαδή η τραπεζική δραστηριότητα στους φορολογικούς παραδείσους. Τουλάχιστον στην Γαλλία μπορέσαμε να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα και πιστεύω πως είναι απαραίτητο να υπάρχει δεν μπορούμε όλα να τα κάνουμε από κοινού, αλλά το να μιλήσουμε για διαχωρισμό δραστηριοτήτων χωρίς να μιλήσουμε για τραπεζικές ε, δραστηριότητες, στους φορολογικούς παραδείσους και τους μηχανισμούς φοροδιαφυγής, τις οποίες, των οποίων χαίρουν οι επενδυτικές τράπεζες θα σήμαινε ότι μιλάμε για ένα βασικό θέμα παραλείποντας ουσιαστικά ε, ζητήματα. Τελικά η πραγματική οικονομία σήμερα ε, αναπτύσσεται και με μέσα, με άμεσες επαφές και, και, και το σύνολο του τραπεζικού συστήματος μέσα στην περιπλοκότητά του έχει εγκαταλείψει μια από τις βασικές δραστηριότητες του που είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και γι' αυτό θα πρέπει να διατηρήσουμε υπόψη μας ότι ο στόχος είναι βέβαια να αυξηθεί η σταθερότητα του συστήματος αλλά επίσης να διατηρηθεί και ο στόχος επιστροφή στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας ε, και να συμφωνήσουμε για ένα σημείο πολύ σημαντικό, όπως το βλέπω τουλάχιστον στην Γαλλία, ότι δηλαδή τι ακριβώς είναι μια δραστηριότητα στήριξης της αγοράς. Είναι ένα θέμα, το είδαμε στην έκθεση του κ. Λάγκερ, όπου πολλά μπορούμε να πούμε και που επιτρέπει κάποιες φορές να εισάγουμε θέματα τα οποία θα είχαμε θελήσει να ε, απομακρύνουμε. Επειδή δεν έχουμε χρόνο και θέλω να απαντήσω σε κάποια από αυτά που είπατε, θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν ε, αν έχει ιδέα για το ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή της νομοθετικής πρότασης και αν μπορείτε αυτό να το κάνετε σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς στοχεύουμε να καταθέσουμε την πρότασή μας ε, το καλοκαίρι. So, aiming, when, when you use the word aiming. <laughs> δηλαδή, τι εννοείται ακριβώς. Achieving that before the summer. Πόσο πιθανό είναι να το πετύχετε αυτό το στόχο. Ναι, αυτό το καλοκαίρι εννοούσα. Το φετινό. Τι θα πει γύρω στο καλοκαίρι. Okay. Κοιτάξτε, κάτι καινούργιο εδώ στο χρονοδιάγραμμά μας είναι ότι τώρα υπάρχει έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας από το Ευρωπαϊκό λέει, Κοινοβούλιο που η Κομισιόν φυσικά θα την προσέξει όλος ιδιαιτέρως αλλά δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένες ενδείξεις τι θα πει καλοκαίρι γιατί οι οδηγίες που έχουμε, οι εντολές που έχουμε από την ιεραρχία μας είναι όσο το δυνατόν συντομότερα το καλοκαίρι. Καλά. Εμεί είμαστε ευέλικτοι και δεν φοβόμαστε τη δουλειά. Μπορούμε να τα δούμε τα πράγματα και διαδοχικά και ταυτόχρονα. Λοιπόν, Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα όσα ελέγχθησαν, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ακούστηκαν εξαιρετικά πράγματα. Για οποιαδήποτε έκθεση βέβαια, ο εισηγητής έχει ορισμένους περιορισμούς στο μήκος που μπορεί να γράψει και εξαρτώμαι από τους σκιώδεις μου να μου καταθέσουν τροπολογίες για να βελτιώσουν τη διατύπωση. Πρέπει ίσως να ξαναδούμε αν είναι όντως υποχρεωτικό να είναι τόσο σύντομες οι εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας ιδιαίτερα για σημαντικά θέματα. Με εντυπωσίασαν μερικά από αυτά που είπατε και νομίζω ότι πρέπει όντως να δούμε τα πράγματα υπό το πρίσμα της αλλαγής νατραπίας γιατί αν περιμένουμε να, κάνει προτάσεις, ε, να κάνουν προτάσεις οι ίδιες οι τράπεζες, η λεγόμενη βιομηχανία δηλαδή, τότε ποτέ δεν θα γίνουν όλα αυτά. Αλλά επειδή όμως είναι έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας μπορούμε να επιδείξουμε πνεύμα καινοτομία. Δεν μας εμπνευσμεύουν άλλοι περιορισμοί που έχουν οι συνήθεις εκθέσεις. Η κύρια ιδέα που ενδιέφερε τους περισσότερους ήταν ο διαχωρισμός. Αλλά ας επανέλθω στην νοοτροπία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν φανερό ότι και στον τομέα της κανονικής, της λιανικής λεγόμενης τραπεζικής δραστηριότητας υπήρξαν παρατυπίες. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να τον προστατέψουμε και αυτόν γιατί μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η ανάπτυξη, η στήριξη της πραγματικής οικονομίας και αυτά που είπαν όλοι σχεδόν οι συνάδελφοι. Πρέπει να το πούμε ρητά, δεν θα ξαναστηρίξουμε τράπεζες εμείς οι, κατα... οι Και για να επανέλθω πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε εθνικοποιημένη τράπεζα, 82% ανήκει στην κυβέρνηση και χρειάστηκε να πληρώσει φοβερά πρόστιμα. You get into σε σχέση με την ε, κρίση του Λάιμπορ. Πληρώθηκαν λοιπόν πρόστιμα στην κυβέρνηση και εν τη σοφία του ο Γεώργιος Όσμπορν είπε ότι έπρεπε μερικά από αυτά τα πρόστιμα να χρησιμοποιηθούν για την περίθαλψη των στρατιωτών μας που ακροτηριάστηκαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Υπήρξε λοιπόν εδώ μια ανακύκλωση των χρημάτων των φαραλαγουμένων. Άρα εδώ χρειάζεται μια μεταρρύθμιση γιατί όλα αυτά έχουν γίνει ανεξέλεγκτα. Και αυτά μπορούμε να τα πούμε σε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Όσο για τους αριθμούς εμπιστοσύνης των ε, καταναλωτών, βλέπουμε ότι δεν συμφωνούν με τις τράπεζες. Πρέπει βέβαια να κάνουμε μια επιλογή. Η Κορίνη είπε, είτε θα ζητήσουμε ολοκληρωμένη εναρμόνιση της ενιαίας αγοράς και αυτό τι σημαίνει. Ότι και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι Κάνουν λάθος. Θα πούμε στους Βρετανούς δεν είναι σωστό το πρότυπο που ακολουθήσατε ή το βρετανικό πρότυπο στόχευε σε μια τραπεζική δραστηριότητα που είναι από τη φύση της πιο που από τη φύση περιέχει μεγαλύτερη ανάληψη κινδύνου από ότι τα ευρωπαϊκά πτυά αυτά. Ορισμένοι είπαν ναι, αλλά πολλές τράπεζες ήδη λειτουργούν διεθνικά και διαμεθοριακά, άρα δεν τίθεται θέμα τι θα κάνουν οι Γερμανοί και τι οι Γάλλοι μόνοι τους. Είτε θα σχεδιάσουμε δικό μας σύστημα ανάμειξη των υπαρχόντων, είτε θα πούμε ότι καθορίζουμε ένα μίνιμουμ κριτηρίων, αλλά που μπορούν και να ξεπεραστούν, είτε θα ξεπεράσουμε και αυτά που προβλέπει η ενιαία αγορά. Πρέπει να τα ξεφθούμε λοιπόν όλα αυτά προσεκτικά. Μ' άρεσαν και άλλες ιδέες που ακούστηκαν για το, την ευθύνη των διευθυντών των τραπεζών και η Σάρον είχε πει ότι στις Ηνωμένε Πολιτείες προσπάθησαν να κάνουν τους σχετικούς ορισμούς και δεν κατέληξαν πουθενά. Δεν είναι το αμερικανικό λοιπόν πρότυπο το καλύτερο. Πρέπει να ξέρουμε τι προστατεύουμε, τι θέλουμε να προστατεύσουμε. Πρέπει να είμαστε μεν ευέλικτοι, αλλά να μην ξεχάσουμε το βασικό θέμα του πώς θα αλλάξει η ανατραπία, πώς θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα και πώς θα προστατεύσουμε τα προστατευτέα. Οι τράπεζες καταθέσεων, οι καταθέσεις και η διαχείρισή τους είναι η βασική δραστηριότητα των τραπεζών. Δεν θέλουμε μόνο μπαλώματα, αλλά μακροπρόθεσμες και βιώσιμες τραπεζικές λύσεις και πρότυπο τραπεζικής δραστηριότητας. Αλλά βέβαια σε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας δεν μπορούμε να προτείνουμε νομοθεσία, μπορούμε όμως να προτείνουμε καινοτόμες λύσεις. Θα σταματήσω εδώ αν δεν απατώμε. Να σας δώσω το χρονοδιάγραμμα. Θα καταθέσω σχέδιο έκθεσης. Θα το γράψω βέβαια πρώτα πριν το καταθέσω. Βέβαια συνήθως χρειάζονται μερικές εβδομάδες και για τις μεταφράσεις και λοιπά. Εγώ όμως θα το διανύμω μόλις το γράψω. Για όσους διαβάζουν αλλά και κατανοούν την αγγλική μετά θα υποβληθεί, θα εξεταστεί στις 21 Μαρτίου της εισημερίας στην Επιτροπή το σχέδιο και μετά η διορία τροπολογιών λίγη στις 15 Απριλίου, 7 Μαΐου η εξέταση και μετά θα ψηφίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να σεβαστούμε αυτό το χρονοδιάγραμμα για να πάει στην Ολομέλεια πριν τον Ιούλιο οπότε και θα εξετάσει την πρόταση η Κομισιόν. Ευχαριστώ λοιπόν τους συναδέλφους για τη συμβολή τους και θα συνεργαστώ και με τους κοιόδης για να πετύχουμε να καταλήξουμε σε προτάσεις λίγο πιο φιλόδοξες από αυτές που έχουμε ήδη ακούσει. Συνεχίζω λοιπόν ως προεδρεύουσα τώρα με το επόμενο θέμα. Η ετήσια έκθεση για τη φορολογία, πώς θα απελευθερώσουμε το ευρωπαϊκό δυναμικό για την ανάπτυξη. Η συγγήτρια είναι η Νίκο Γκαλπέλς από το ΕΛΚ και θα, το δώσω, θα το δώσω όμως τον λόγο και μετά θα ακούσουμε τους και συγγήτες. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ λέει η κυρία Πέλς, Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Επίσης, λόγω του ότι ε, έχετε λάβει την έκθεση πριν από λίγες εβδομάδες στη μητρική σας γλώσσα. Θα ήθελα λοιπόν να παρα... παρουσιάσω τις αλλαγές στη φορολογική πολιτική στην Ένωση του 2012 με λίγα λόγια να πω πως ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών υιοθετήθηκε, εισήχθη σε 11 κράτη-μέλη και για την περίοδο 2014-2020 ε, υπάρχει ένα σχέδιο δράσης φορολογικής πολιτικής που είναι ένα νομίζω μια καλή κατεύθυνση όπως λέει και ο τίτλος μου στην έκθεση ε, στόχος μας είναι να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό είναι δύσκολο λόγω των ε, αυστηρών ε, ρυθμίσεων που υπάρχουν στα δημοσιονομικά λόγω της κρίσης, αλλά επισημαίνουμε πως υπάρχει μια διάθεση για μια φορολογική πολιτική η οποία θα ευνοεί την ανάπτυξη. Αρκετά κράτη-μέλη έχουν τέτοιες πολιτικές, αλλά θεωρώ πως πρέπει να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις πολιτικές για να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας η φορολογική πολιτική. Πρέπει να έχουμε έξυπνους φόρους στην κατανάλωση αντί για την παραγωγή έτσι ώστε το διαθέσιμο εισόδημα να διοχετεύεται στις αποταμιεύσεις. Επίσης σημαντικό είναι να σημειώσουμε πως ε, υπάρχουν τρεις παραγωγικοί τρεις παράγοντες παραγωγής η εργασία, το κεφάλαιο και η τεχνολογική πρόοδος και εκεί πρέπει να κινηθεί και η φορολογία επιπλέον η φορολογική πολιτική μπορεί να ακολουθήσει ένα μοντέλο δύο φάσεων για να αναζωογονήσει την οικονομία και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη ε, ζήτηση για να οδηγήσουμε έτσι και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Όσον αφορά τώρα το ποσοστό, το ύψος του φόρου και τους νέους φόρους, νομίζω πως καλύτερο είναι μεταξύ των δύο να διευρύνουμε την υφιστάμενη φορολογική βάση για περισσότερα έσοδα. Είναι καινοτομία του σχεδίου αυτού πως παρά το ότι σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, εισάγει το λεγόμενο φορολογικό φίδι. Αντί... Αντί λοιπόν για εναρμόνιση λαμβάνονται υπόψη ε, οι περικοπές των φόρων και το πάγωμα των φόρων στα κράτη-μέλη για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των κρατών μελών και βεβαίω, όπως ξέρετε επειδή υπάρχει περιορισμός λέξεων δεν μπόρεσα να αναφερθώ στα μέτρα καταπολέμησης φορολογικής απάτης αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε αλλά όπως τονίστηκε και στο φορολογικό πρόγραμμα του ΩΣΑ για το 2012 πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ε, επιθετικές φορολογικές πολιτικές των εταιριών και την κατάχρηση των ε, φορολογικών παραδείσων. Η διαφάνεια των φορολογικών καθιστώτων είναι απαραίτητη γιατί αλλιώς υπάρχουν ε, απώλειες δισεκατομμυρίων στους προπολογισμού των κρατών μελών. Και αν δεν καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο θα ενισχυθεί η μαύρη οικονομία και θα υποβαθμιστεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών και την φορο συλλεκτική ικανότητα γιατί θα μειωθούν και τα δημόσια χρέη και είναι αναπόφευκτο τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τη συνεργασία των φορολογικών διοικήσεων. Είναι επίσης αναγκαίο η Κομισιόν να δημοσιεύσει τους μηχανισμούς παρακολούθησης των μέτρων και την βαθμολογία σας ευχαριστώ λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι. Έχετε το σχέδιο έκθεσης και αναμένω τα σχόλια ε, και από τους συνάδελφους και τους κοιόδης εισηγητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια Όλε Λουντβίχισεν τώρα για τους σοσιαλδημοκράτες. Να ευχαριστήσω καταρχήν την εισηγήτρια για την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση είναι ενδιαφέρουσα διότι εστιάζει στη σύνδεση ανάμεσα, στη σχέση ανάμεσα στις ε, φόρους και τις, την ανάπτυξη. Είναι μια πολύ σημαντική πτυχή αυτή, περισσότερο από ποτέ, αλλά δυστυχώς συχνά παραμελείται. Πρέπει να σκεφτούμε τρεις βασικές αρχές. Καταρχήν, είναι απαραίτητο να εντατικοποιηθεί η εθνική και η ευρωπαϊκή προσπάθεια όσον αφορά την φοροδιαφυγή και τις φοροαπάτες. Ξέρουμε ότι η Κομισιόν του τελευταίους έξι μήνες έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό και τώρα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτά όλα θα μετατραπούν σε συγκεκριμένες δράσεις. Ε, Επίσης ε, θα πρέπει να υπάρξουν ευνοϊκές ε, συνθήκες για βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και αν θέλουμε να έχουμε πιο ε, δίκαιους και πιο ισότιμους κανόνες ανταγωνισμού δεν υπάρχει λόγος τότε να προσπαθεί κανείς να αποφύγει το σύστημα ή να φοροδιαφύγει. Ίσως ε, βέβαια θα πρέπει να εξετάσουμε και την κοινωνική πτυχή εδώ και θα ήθελα αυτό να αντιμετωπίζεται στην έκθεση ότι δηλαδή δεν θα πρέπει να έχουμε τέτοια φορολογική δομή που να αυξάνει το σε διακρίσεις στην κοινωνία. Αυτή, αυτά τα ευρύτερα ε, κενά είναι απαράδεκτα και επηρεάζουν την ανάπτυξη. Περισσότερα κράτη-μέλη αυξάνουν τους φόρους στην κατανάλωση αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και διευρύνει το κοινωνικά τις κοινωνικές αποκλήσεις. Ε, γιατί αυτό σημαίνει πως ε, κάποια από τα πιο χαμηλά, χαμηλόμιστα νοικοκυριά πρέπει να πληρώσουν περισσότερους ε, φόρους αναλογικά και γι' αυτό και θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Και όσον αφορά την, τους φόρους κατανάλωσης, ε, αυτό δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι η προοδευτικότητα στα φορολογικά συστήματα θα υποβαθμίζεται. Η περιβαλλοντική ιδέα νομοθεσία είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της ανάπτυξης. Η ιδέα που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι ότι ο περιβαλλοντικός φόρος ε, παρακμάζει και αυτό δεν είναι καλό γιατί για την ανάπτυξη είναι πολύ σημαντικό η περιβαλλοντική νομοθεσία να καλύπτει με καλύτερο κομμάτι της γενικής νομοθεσίας. Το χρειαζόμαστε αυτό για τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και πρέπει να μπορέσουμε να κινηθούμε προς την πράσινη οικονομία και αν θέλουμε αυτό να είναι επιτυχές χρειαζόμαστε περιβαλλοντική νομοθεσία. Επιπλέον χρειάζεται αναθεωρημένη οδηγία περί φορολογίας της ενέργειας με φιλόδοξους στόχους ε, και τέλος είναι δυνατόν να κάνουμε περισσότερα για την ανάπτυξη αφαιρώντας ε, τα φορολογικά εμπόδια που υπάρχουν στην ενιαία αγορά και η προσέγγιση προς την οδηγία για την φορολόγηση θα πρέπει να είναι ότι πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα στην νέα αγορά. Η εξυγίανση του, της βάσης για τον φόρο των επιχειρήσεων μπορεί να απλοποιηθεί αν εφαρμοστεί και σωστά και η συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές φορολογικές αρχές και των διαφόρων κατανομιλών θα πρέπει να γίνεται σωστά στο μέλλον. Δύο μόνο ακόμα παρατηρήσεις έχω να κάνω σε σχέση με το σχέδιο έκθεσης. Το φορολογικό φίδι για να υπάρξει με στόχο το καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στις εθνικές φορολογικές αρχές θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Τι είναι αυτό το φίδι. Ήταν, είναι αυτό όπως το φίδι το οποίο προηγήθηκε του ευρώ. Εάν ναι, και θέλουμε να πάει προς την εναρμόνιση της φορολογίας, πρέπει να το συζητήσουμε. Το διπλό, μάλλον το πρότυπο δυο βημάτων για την εναρμόνιση της φορολογίας, όπως αναφέρεται στην έκθεση, κίνητρα προς τις εξαγωγές και προς την απασχόληση. Θα πρέπει αυτό να τα εξετάσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες, νομίζω. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το κείμενο αυτό. Πολύ καλή αρχή για τη συζήτηση και προσβλέπω στις συζητήσεις μας ε, την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Τώρα δεν έχουμε άλλο χρόνο και δεν ξέρω αν μπορώ να ζητήσω από τους ερμηνείς να μείνουν περισσότερο. Γι' αυτό θέλω να είστε σύντομοι στα σχολεία σας. Εξ ονόματος της ΑΛΤΕ έχουμε τον κύριο Μπαλτέ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μερικά σχόλια. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Είναι καλή εκκίνηση αυτή η εργασία για να αναρωτηθούμε πώς θα μπορούσε η Ευρώπη να βελτιώσει τα πράγματα για την ανάπτυξη και τη φορολογία. Και οι φιλελεύθεροι συνάδελφοί μου και άλλοι θα καταθέσουμε τροπολογίες όπου θα μιλούμε για την ανάγκη εφαρμογής μεταρρυθμίσεων, όχι μόνο περιορισμούς και περικοπές, να μην ξεχάσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Μπορούμε να μιλήσουμε φυσικά για αύξηση φορολόγηση. Εγώ είμαι υπέρ του φόρου των δοσοληψιών, ας πούμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα τον προϋπολογισμό ως προϋπόθεση. Στις Ηνωμένε Πολιτείες μετά από μερικά χρόνια και ενσιανισμού βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα για να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται και που θα δημιουργήσουν την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Επίσης, σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες είδαμε ότι περικόπτουν τις δημόσιες δαπάνες αλλά αν παραμείνουν μονοπόλια και γραφειοκρατίες και αν η αγορά εργασίας συνεχίζει να μην είναι ελαστική δεν θα αποδώσουν όλα αυτά. Δεύτερον, αυτά όλα ήταν το πρώτο. Δεύτερον, είμαι υπέρ της, του φορολογικού ανταγωνισμού. Είναι πολύ φιλελεύθερη ιδέα βέβαια, αλλά πρέπει να, τον διατηρήσουμε. Έχουμε κοινό νόμισμα, κοινή νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη, αλλά πρέπει να εναρμονίσουμε την βάση της φορολόγησης των επιχειρήσεων τουλάχιστον, όχι όμως μόνο. Χρειάζεται ανταγωνιστικότητα που θα ήταν καλή για όλες τις οικονομίες και θα καταθέσουμε τροπολογίες σχετικώς. Η αμερικανική εμπειρία νομίζω είναι θετική, αλλά η φορολογική ε, όχι και τόσο. Πρέπει να γίνουν διορθώσεις για να μπορέσει να προσαρμοστεί κάθε χώρα με τη διαφορετική πολιτική που ασκούν οι άλλες. Αυτό που εναρμονίζουν οι Αμερικανοί είναι τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και της αγοράς εργασίας. Αυτό δεν το έχουμε στην Ευρώπη. Ας πούμε υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες διαφορές στην Ευρώπη μεταξύ της αγοράς εργασίας της Δανίας και της Ισπανίας, παραδείγματος χάρη. Μεγαλύτερη από ό,τι στις διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων. Αυτό είναι που κάνει την Αμερικανική οικονομία πιο αποτελεσματική. Τέλος, για τη φορολογική εξαπάτηση πρέπει να εφαρμόσουμε τις βέλτικες πρακτικές των καλύτερων ευρωπαϊκών χωρών και να βασιστούμε στα στατιστικά στοιχεία των χωρών που έχουν τη μικρότερη φοροδιαφυγή. Αυτές είναι οι μικρότερες βέβαια. Ευέβητα οι μικροφορολογικές απάτες ή οι φορολογικές μικροαπάτες σημειώνονται σε μοσπονδιακές χώρες όπως τη Γερμανία όπου 17 οντότητες συλλέγουν τους φόρους. Έτσι μειώνονται οι απάτες. Στην Ισπανία δύο περιοχές, η Ναβάρα και η Βασκία, συλλέγουν μόνες τους τους φόρους τους και εκεί σημειώνονται λιγότερες απάτες. Νομίζω λοιπόν ότι όσο μεγαλύτερο είναι η επικράτεια της συλλογή των φόρων, Τόσο ε, περισσότερες και μεγαλύτερες είναι και οι φορολογικές απάτες. Σας ζήτησα να είστε και λίγο σύντομοι, γιατί ο χρόνος μας έχει δει τελειώσει. Φιλίπ, εγώ θα διαφωνήσω, Ραμόν. Γιατί ως πολίτης, όταν έχουμε φορολογικό ανταγωνισμό, ποιος κερδίζει. Ποιος κερδίζει. Οι μεγάλοι μεγάλες εταιρείες και ως φιλελεύθερος δεν θέλεις φαντάζομαι οι μεγάλες εταιρείες να έχουν αθέμητα πλέον εκτήματα γιατί θέλεις ανταγωνισμό και οι μεγάλοι όταν μιλάμε για το, για το ατομικό εισόδημα. Οπότε δεν θέμε να χαλαρώσουν οι κυβερνήσεις και να θεωρούν πως δεν υπάρχει λόγος να είναι αποτελεσματικές, οπότε πράγματι πρέπει να ασκηθεί κάποια πίεση. Και ως ένα βαθμό θα σκεφτεί κανείς πως νέο ανταγωνισμός δημιουργεί αυτή την πίεση. Δεν λέω λοιπόν να χαλαρώσουμε κάθε πίεση. Αυτό το οποίο λέω είναι ο αχαλήνοτος ανταγωνισμός κάνει τους μεγάλους να μην πληρώνουν και καταλήγουν να πληρώνουν οι μικροί. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσει πληρώνουν πλήρω. οι μεγάλες δεν το κάνουν. Δείτε την ε, έκθεση πριν από δύο... την έκθεση, με συγχωρείτε, που πριν από δύο εβδομάδες. Πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε συγκεκριμένα τον τομέα της φορολόγησης των επιχειρήσεων ως ένα τομέα που πρέπει να γίνει περισσότερα, να υπάρξει κοινή ενιαία φορολογική βάση. Όχι όμως με ένα ύψο ύψος φορολογίας, αλλά για καλύτερη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Βεβαίως δεν θα σε καταπλήξει το ότι οι πράσινοι επιμένουν πως πρέπει να φροντίσουμε η φορολογία να χρησιμοποιείται και για να ενσωματώσει τις περιβαλλοντικές εξωτερικότητες οι οποίες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις τιμές αγοράς και άρα να προωθήσει την Κομισιόν για περαιτέρω φορολόγηση της ενέργειας και το Συμβούλιο. Και αυτό είναι το ελάχιστο για εμάς. Θα σταματήσω εδώ. Ενδιαφέρουσα συζήτηση και δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς να τη συνεχίσουμε. Θα το ξαναδούμε στις στη συζήτηση των τροπολογιών. Ο κ. Σίτσεκ για τους Ευρωπαίου Συντηρητικού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ε, και ο χρόνος έχει τελειώσει. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος κι εγώ. εσεί τουλάχιστον ως Πρόεδρος και η κυρία Σιγήτρια θα θυμάστε την παρατήρησή μου της προηγούμενης εβδομάδας ε, για μια άλλη έκθεση για τα φορολογικά και χαίρομαι πως για το ότι και αυτή η έκθεση είναι ε, πάρα πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Είναι οργανωμένη σωστά σε τρία τμήματα. Το πρώτο μέρος τώρα. Το πρώτο μέρος δεν έχω κάποιες φοβερές αντιρρήσεις και χαίρομαι και για την διατύπωση η οποία βασίζεται σε μια οικονομική φιλοσοφία με την οποία σχεδόν ε, ταυτίζομαι. Στο δεύτερο μέρος, θετικό είναι το κομμάτι όπου μιλάτε για τις νέους πόρους. Και εκεί πέρα έχετε χαμηλό προφίλ, δεν μιλάτε ούτε για επιπλέον πόρους, ούτε για αυξήσεις ε, φόρων, με το οποίο συμφωνώ. Και συμφωνώ για να ξεκαθαριστεί και αυτό, με την θέση πως πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φορολογική απάτη καλύτερα, αντί να αναζητούμε νέους πόρους. Η συζήτηση με τον Φιλίπ για τους περιβαλλοντικούς φόρους τώρα αναβάλλεται. Και να σας διαβεβαιώσω, κυρία εισηγήτρια, πως ε, θα υποβάλω τροπολογίες αλλά κατά την άποψή μου δεν θα σας δυσκολέψουν πολύ. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε. Κυρία Σίγητρε, ευχαριστώ σύντομα. Θα ήθελα και εγώ να απαντήσω itt is köszönöm mindenkinek az észrevételét és javaslatát. E, ami ευχαριστώ για όλα σας τα σχόλια. Δείχνουν πως αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα που αναφέρατε. Οπότε μπορούμε είτε να δούμε όλη τη διαδικασία είτε να τη δούμε κομμάτι-κομμάτι. Το πρόβλημα, όπως το βλέπω εγώ, είναι πως έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες και δεν κάνουμε τίποτα. Η μέθοδος που θα ήθελα να ακολουθήσω και ζητώ εδώ τη στήριξή σας είναι να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα, μικρά βήματα που μπορούμε να υλοποιήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη. Από κοινού σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για τη μέθοδο. Υπάρχουν κάποια βασικά πράγματα που ήθελα να μείνουν στην έκθεση. Σε κάποια άλλα βεβαίως δέχομαι τροπολογίες. Δεν συμφωνώ πλήρω με όλες τις απόψεις που ακούστηκαν βεβαίως. Ναι, νομίζω πως έχουμε πολλές ευκαιρίες σε επόμενες συναντήσεις να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Επίσης θα ήθελα να ε, εξηγήσω την ιδέα του φορολογικού φιδιού που είναι μια καινοτομία. Επίσης να δεχτώ μια κοινωνική προοπτική, αλλά μη γίνει τώρα το ζήτημα κοινωνικών φόρων το κύριο σημείο της έκθεσης. Πρέπει να διαχωριστούν αυτά τα κείμενα, τα θέματα στο κείμενο. Για το περιβάλλον είχα βάλει κάτι και το έβγαλα. Δύο φορές γιατί είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι αυτή η έκθεση το κατάλληλο σημείο. Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή και η απάτη. Και αυτά τα βγάλα γιατί υπάρχει άλλη έκθεση μετά που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Για το φορολογικό ανταγωνισμό τώρα και το ποιος κερδίζει είναι θέμα οικονομικής θεωρίας που και πάλι δεν νομίζω πως πρέπει να απασχολήσει την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις και θα ήθελα να τονίσω πως η προθεσμία των τροπολογιών είναι η 5η Μαρτίου και εγώ θα ήθελα να καταθέσω τις τροπολογίες γιατί υπήρχαν κάποια ζητήματα που δεν μπόρεσα να τονίσω στην έκθεση και στις 5 Μαρτίου θα ήθελα να συναντηθούμε δύο με 3 το απόγευμα θα αποστείλω προσκλήσεις. 5 Μαρτίου, μάλιστα, 11 Απριλίου θα δούμε τις τροπολογίες, θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή 24 Απριλίου για να πάμε στην Ολομέλεια του Μαΐου. Και θα συναντηθείτε με τους ηγητέ ε, στο Στρασβούργο. Δεν υπάρχει τίποτα στα διάφορα. Η επόμενη συνεδρίαση στο Στρασβούργο, Δευτέρα 11 Μαρτίου, 7 το απόγευμα. Ευχαριστώ, γεια σας.